Ladies and gentlemen, it's now 2.30 and um, uh, you were going to have the fun of myself in this chair this afternoon. In fact, uh, the chairman who I see is now arriving. Έρχεται τώρα ο πρόεδρος, λίγο νωρίτερα από ό,τι περίμενα. Μου είχε ζητήσει να κάνω το συντονιστή σήμερα το απόγευμα και να πηγαίνω αριστερά και δεξιά και να σας λέω τι πρέπει να κάνετε. Αλλά ήρθε ο ίδιος ο πρόεδρος και θα καθίσει και πρέπει λοιπόν να εκενώσω τη θέση του. colleagues because uh, Mr. Kirkhove had kindly. ο κύριος Κύρκο άρχισε τη συνεδρίαση ήδη, δεν θέλω να διακόψω κι εγώ. το είχα ζητήσει για ένα μισάωρο, όχι ότι πήγε να με ρίξει από την καρέκλα και να κάνει επανάσταση, του είπα εγώ να με αντικαταστήσει μισή ώρα γιατί είχαμε τη συνέντευξη τύπου για την υπουργική. Αλλά τελείωσε εγκαίρος και ήρθα και εγώ εγκαίρος. Θέλω να τον ευχαριστήσω και πάλι που ανέλαβε. Ε, και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω. Δεν είναι και η πρώτη φορά που με διευκολύνει. Με έχει βοηθήσει και εμένα και τη γραμματεία και στο παρελθόν. Τίμω, ευχαριστώ. Και όντω ε, σου άρεσε ε, να κάθεσαι στην καρέκλα μου, το είδα. Λοιπόν, ε, σημεία 6, 7 και 8 πρέπει να αναβληθούν ε, διότι... Εγώ είμαι της, διότι δεν έχουμε τις γνωμοδοτήσεις από την νομική υπηρεσία. Εάν δεν έχετε αντιρρήσεις, θα εγκριθεί έτσι η μερίσια διάταξη. Okay. So just go on to the endorsement of coordinators' Θα ήθελα λοιπόν βάσει του κανόνα 205 του ιστορικού κανονισμού να διεκπαιρεώσω το ταχύτερο δυνατόν κάποια σημεία για το διορισμό των εισηγητών. Έχουμε τη Μόνικα Χολμαϊέρα από το ΕΛΚ για την ε, ε, έκθεση ε, της οδηγίας 2011-93 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης των παιδιών. Επίσης έχουμε διορισμούς εισηγητών, είναι αρκετά σημαντική και γι' αυτό παρακαλώ προσέξτε με να σας πω. Η Σκά Κέλλερ από τους Πράσινους για πρόταση για την απόφαση του Συμβουλίου για τη θεσπίση μέτρων για τη διεθνή προστασία για την Ιταλία και την Ελλάδα, ο μηχανισμός ανάκλησης δηλαδή. Στη συνέχεια διορισμού εισηγητή για μία γνωμοδότηση ο κύριος Πίτερ Νίντερ Μίλλερ από τους σοσιαλιστές για την ε, κινητοποίηση των ε, ε, οργάνων ευελιξίας για τα προσωρινά μέτρα στον τομέα πάλι της διεθνούς προστασίας για την Ιταλία και την Ελλάδα. Επίσης, οι συντονιστές στην τελευταία του σύσκεψη συμφώνησαν και για μελλοντικές ημερομηνίες συνεδριάσεων. Είναι λεπτό το ζήτημα αυτές οι επιπρόσθετες συνεδριάσεις, αλλά χρειαζόταν ε, γιατί θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι εξαιρετικά μεγάλος ο φόρτος εργασίας. 5η ε, 2 Ιουλίου το απόγευμα στη, στο Στρασβούργο ε, στις 7 το βράδυ, 6 Ιουλίου στο Στρασβούργο με τον Επίτροπο Αβραμόπουλο και την ε, είπατε εκπρόσωπο Μογκερίνη για την στρατηγική έκθεση ε, για τη μετανάστευση. Δευτέρα στο Στρασβούργο, έτσι. Τώρα η κατάσταση για τα ΜΜΕ στη Σλοβακία, βάλει οι συντονιστέ το ζήτησαν μετά από την, κυβέρνηση, την απόφαση τη κυβέρνηση τη Σλοβακία να απαγορεύσει την επικοινωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση και την ε, εφημερίδα NDENK ζήτησαν ε, οι συντονιστέ από μένα να γράψω μια επιστολή προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την καλύτερη νομοθεσία, οι συντονιστέ ε, συνέστησαν να γράψουμε μια επιστολή στον πρόεδρο Σούλτ με τι προτεραιότητε τη ΛΥΜΠΕ σε σχέση με την αθέρωση των κανόνων για την καλύτερη νομοθεσία. Αποστολέ. Παρακαλώ προσέξτε με συναδελφοί αν έχετε δηλώσει και συμμετοχή στις αποστολές ε, Φινλανδία για το πακέτο ε, ευθείων συνόρων ε, τρία μέλη και όχι τέσσερα, όπως είχαμε λάβει την έγκριση. Θα έχουμε ένα βουλευτή από το ΕΛΚ και ένα από τους σοσιαλιστές που θα καλύπτουν δηλαδή, τους δύο εισηγητές και έναν βουλευτή από το ECR. Για την Σικελία αποφάσισαν οι συντονιστές ότι πρέπει να στείλουμε έξι μέλη της Επιτροπής και με την επιπρόσθετη δυνατότητα να υπάρχουν και συνοδευτικά μέλη από την Ιταλία Στη συνέχεια έχουμε το, το φόρουμ της διακυβέρνησης του Διεδικτύου 2015 στην Βραζιλία. Θα ζητήσουμε σύνδεση για την αποστολή μας και θα γράψουμε επιστολή προς τις Επιτροπές Ιτρεκάλτζουρι και ΣΤΟΑ. Ε, στη συνέχεια για τα, τις προτάσεις ψηφισμάτων κανόνας 133 θεώρησαν οι συντονιστές ότι δεν χρειάζεται follow-up και σας απαριθμώ για, ε, για ποιες προτάσεις μιλάμε. Β80497 2015 για την παρενοχληση στοκιν στόκινγκ Β80498 για την αναγνώριση της σημασίας ε, του ρόλου και του έργου των αστυνομικών δυνάμεων ε, Β80486 2015 για την Ευρωπαϊκή Συγγελία για την Καταπολέμηση της Τρομοκράτειας, Β80519-2015 για την κατάσχεση εγαθών που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητε και τέλος Β80488 για έργα τέχνης που έχει καταστρέψει το Ισλαμικό κράτος. Μετά περνάω τώρα στην επιστολή που στείλαμε στην Επιτροπή Αναφορών από, σχετικά με την αναφορά του Ντάνιελ Πένια Ζορτάνα από τον Frontex σε σχέση με την αύξηση, διεύρυνση μάλλον των αρμοδιοτήτων και την αύξηση της χρηματοδότησης. Βάσει του κανόνα 205 μπορείτε να εγκρίνετε τι στάσεις των συντονιστών. Ωραία, εγκρίθηκαν πολύ ωραία. Και μετά από αυτές τις παρατηρήσεις μπορείτε να ελέγξετε αν έχετε έτοιμες τις κάρτες σας γιατί στις 4 και 20 θα ψηφίσουμε. Είναι σύντομη αλλά πολύ σημαντική ψηφοφορία και παρακαλώ να φροντίσετε να τις έχετε τι κάρτες σας. 4 και 20. Πάμε τώρα στο σημείο 4 της σε διαταξής ε, είναι η πρόληψη ριζοσπαστικοποίησης και στρατολόγησης Ευρωπαίων πολιτών από τρομοκρατικές οργανώσεις της Ρασίτα Ντατή. Θα εξετάσουμε το σχέδιο έκθεσης. Ξέρετε πόσο σημαντικό και πολύ σύνθετο είναι αυτό το θέμα, συνάδελφοι. Στη ΛΥΜΠΕ έχουμε κάνει διάφορες συζητήσεις για αυτό το θέμα. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση θα δώσω το λόγο στην εισηγήτριά μας για την παρουσία του σχεδίου έκθεση. Κύριε Ντατή. Ευχαριστώ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς θα είμαι πολύ σύντομη, διότι αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι να συζητήσουμε και να ακούσουμε τις προτάσεις και τις απόψεις όλων των μελών της Επιτροπής αυτής. Σας έστειλα το σχέδιο εκθέσεως όσον αφορά τη ριζοσπαστικοποίηση και την, τοστατολόγηση Ευρωπαίων πολιτών από τους τρομοκράτες. Ε, συμμετείχα στη σύνταξη λοιπόν του κειμένου, προσπάθησα να λάβω υπόψη όλους τους τομείς που, και τους τόπους που να δράσουμε για να πετύχουμε το στόχο. Αυτό που είδα από τι ακροάσεις και τι συναντήσει ότι όλοι ζητούν μια στρατηγική σφαιρική για την πρόληψη τη ριζοσπαστικοποίηση στην Ευρώπη. Κάθε χώρα αναφέροντα ότι δεν μπορούμε ο καθένα να κινηθεί μόνο του ή να λάβει μέτρα απομονωμένα ο καθένα στη χώρα του και να αντιδρά κάθε χώρα συναρτήσει ε, αποπειρών γεγονότων, σοβαρών γεγονότων που συμβαίνουν στη χώρα. Όσον αφορά τη Γαλλία, μετά τις, ε, τα γεγονότα του Ιανουαρίου είδα ότι μετά τις ακροάσεις έχει καθυστερήσει πολύ η Γαλλία όσον αφορά την πρόληψη της ρίζος σε σχέση με τη Δανία, τη Βρετανία ή και το Βέλγιο. Η στατηγική σε ευρωπαϊκό επίπεδο σφαιρική είναι κάτι απαραίτητο. Τώρα ε, διερωτήθηκα για κάποια σημεία όπως πώς να προβλέψουμε παρά να αντιδρούμε στη ριζοσπαστικοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών και όταν ταξίδευα για τις ακροάσεις είδα ότι τα βασικά ε, τα στοιχεία της ριζοσπαστικοποίησης ανεξάρτητα τη χώρα, την περιοχή είναι κάτι που γίνεται μέσω διαδικτύου και πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να το παραδεχτούμε ότι από εκεί γίνεται. Και μπορούμε να το συζητήσουμε το θέμα του δικτύου. Το διαδίκτυο λέγω έγινε ένα σημείο εικονικό εκπαίδευσης πολλών ατόμων που θέλουν να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Και δεύτερος τόπος ριζοσπαστικοποίησης είναι άτομα ε, που είναι ε, στη φυλακή που στατολογούνται. Εκτείουν την ποινή τους και αυτοί που είναι καταδικασμένοι για τρομοκρατία βρίσκονται επιμακρό στη φυλακή. Και εκείνοι που, εκείνοι που τελικά υποκύπτουν είναι αυτοί που είναι κατάδικοι κοινού δικαίου και έχουν μικρές πίνες. Δεν τους εντοπίζουμε, ριζοσπαστικοποιούνται και μετά βγαίνουν σαν ε, βόμβα με θριαλίδα. Λοιπόν, ε, συνάντησα διάφορους ανθρώπου συζήτησα συζήτησα και του παρόχου υπηρεσιών στο διαδίκτυο. Θεωρώ ότι είναι αφελεί οι πάροχοι. Έχουν και διακυβεύματα οικονομικά και κέρδη και δεν είναι πρόσημοι να, να κινηθούν. Τα αιτήματά μας να διαγράψουν τα κείμενα που την τρομοκρατία ή να προβάλλουν τα αντιπιχειρήματα όσον αφορά το θέμα αυτό. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Δεν μπορούμε το διαδίκτυο να υποκρίνεται ότι τίποτα δεν συμβαίνει δεν είναι ένας ολίνας που είναι φορέας ε, διαδόσεως ε, μηνυμάτων τέτοιων, παρακινώντας προς την ριζοσπαστικοποίηση και την τρομοκρατία και τη μυσαλλοδοξία. Όμως είναι μια πραγματικότητα και δεν θα πρέπει να παραμείνουμε αδρανείς. Ε, θα στείλω σχετικά μια επιστολή προς τους υπευθύνους του διαδικτύου όσον αφορά τη φυλακή. Συνάντησα λοιπόν σε φυλακές και είδα κάποια πειράματα που έγιναν εκεί. Όλο το σοφρονιστικό προσωπικό στη Γαλλία και τη Βρετανία ζητούν κατάρτιση γιατί παραμένουν θεατές του φαινομένου αυτού της ριζοσπαστικοποίηση Βλέπουμε αλλαγή συμπεριφορά των ανθρώπων ε, που έρχονται σε επαφή με άτομα ριζοσπαστικά ή καταδικασμένα για τρομοκρατία ή για απόπειρε και αυτά τα άτομα που είναι εκεί για δικήματα του κοινού δικαίου, κάπου χαμένα άτομα, ξαφνικά σαν πρόσχημα παίρνουν τη θρησκεία για να ριζοσπαστικοποιηθούν. Ε, υπάρχουν και διάφοροι μουσουλμάνοι που ασχολούνται ε, με την ελεημοσύνη και λοιπά και τη βοήθεια ε, και δεν στέφονται προς τα... Και αυτοί λένε οι ιερείς ότι δεν έρχονται προς εμάς γιατί λένε ότι είμαστε κακοί οι μουσουλμάνοι. Θα πρέπει λοιπόν να διευρύνουμε όλες αυτές τις δοκιμές και τους πειραματισμούς που γίνονται και τις πληροφορίες που συλλέγονται στις φυλακές για να μπορούμε να παρατηρούμε, να εντοπίζουμε τα άτομα που κάνουν αυτό τον προσλητισμό. Αλλά το σοφρονιστικό προσωπικό έχει πολλές πληροφορίες όσον αφορά τις διαδικασίες που ακολουθούνται για τη ριζοσπαστικοποίηση, αλλά δεν γνωρίζουν πώς να αναλύσουν την πληροφορία, δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση. Ζητή το προσωπικό, την κατάρτιση, για να μπορεί να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες και να τις δώσει σε εκείνους που θα μπορούν να συμβάλλουν να αποφευθεί η ριζοσπαστικοποίηση ή να μην βγουν από τη φυλακή και να μπορούν να κινούνται ελεύθερα εξαιρετικά επικίνδυνα άτομα. Μια άλλη μία μελιτέα πτυχή. Ο ρόλος της παιδείας, της ε, ένταξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο Λέγαμε το αγγλικό, το γαλλικό, το γερμανικό μοντέλο, ο καθένα είχε μοντέλο. Σήμερα έγινε η ένταξη αυτή, ευρωπαϊκό θέμα, αφορά τους Ευρωπαίους πολίτες. Όσον αφορά την παιδεία και την ένταξη, αυτό είναι ένα θέμα που αφορά μια στρατηγική που θα έπρεπε να έχουμε, ευρωπαϊκή στρατηγική, που θα αφορά την ένταξη και την παιδεία. Δεύτερο θέμα και ερώτηση όταν τα μέτρα της πρόληψης απέτυχαν όσον αφορά τη ριζοσπαστικοποίηση, πώς αποφεύγουμε τη στατολόγηση και την αναχώρηση των Ευρωπαίων πολιτών και προφανώς την επιστροφή. Συστήσαμε να υπάρχει συστηματικό έλεγχο, να μην πω συστηματικό, στα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω των Ευρωπαίων πολιτών, διότι σήμερα οι περισσότεροι τζιχαντιστέ και αυτοί οι ξένοι μαχητέ είναι ξένοι μαχητέ για του τόπου του πολέμου, αλλά όχι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν συναντήσετε τους υπευθύνους των αρχών του Ιράκ ή στη Συρία, τη Συρία ή το Αφγανιστάν, μας λένε υπεύθυνοι, κοιτάξτε μπορείτε να συγκρατήσετε τους πολίτες σας που έρχονται να αποσταθεροποιήσουν τη μάχη μας κατά των τζιχαντιστών και κατά του Ισλαμικού κράτους. Οι Ευρωπαίοι πολίτες που αναχωρούν προς αυτές τις χώρες θα πρέπει όταν επιστρέφουν αυτοί να μπορούμε να τους ελέγξουμε και να γνωρίζουμε πότε επέστρεψαν επί της Ευρωπαϊκής Επικράτειας. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα και το συζήτησα εκτενώς με την ομάδα των Πρασίνων περισσότερο, καλύτερη συνεργασία όσον αφορά τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει άμεση χρηματοδότηση ε, των τρομοκρατών από κάποια χώρα. Αλλιώ θα ήταν πολύ εύκολο. Θα ξεκινούσαμε κάποιε διαδικασίε κατά κάποιε χώρε που είχαμε αποδείξει ότι άμεσα χρηματοδοτεί τρομοκρατία. Αλλά δεν είναι τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα, είναι πιο πονηρά τα μέτρα. Στην υποσαχάρη Αφρική υπάρχουν πολλά χρήματα προέρχονται από κάποιες χώρες συγκεκριμένες που χρηματοδοτούν ε, κάποιες σχολές του κορα, κορανικές και ε, λένε εμείς θα δώσουμε παιδεία στα παιδιά γιατί δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο και χρηματοδοτούν ενώσεις, δομές, σχολεία αυτές οι χώρες και σε αυτά τα μέρη, στους χώρους γίνεται ριζοσπαστικοποίηση μέσω του σαλαφισμού κυρίως στις χώρες υποσαχάριας Αφρικής και αυτά τα άτομα ριζοσπαστικοποιούνται και το είδαμε άλλωστε αυτό στην υποσαχάρια Αφρική όταν είχαμε τα, τα σκίτσα του Μωάμετ σε κάποιες εφημερίδες πως σε κάποιες αφρικανικές χώρες είδαμε εμφυλίους πολέμους σε κάποιες περιοχές και αυτά τα άτομα πολύ συχνά ευνοήθηκαν από χρηματοδότηση ή από εκπαίδευση σε αυτές τις δομές που χρηματοδοτούνται κυρίως από τις χώρες του κόλπου. Πρέπει να το πούμε αυτό. Εγώ έγραψα στις χώρες που αποτελούν το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου να τους ε, ζητήσω να είναι πολύ πιο ε, δραστήριοι και να συμμετέχουν στις προσπάθειες η χνηλασιμότητα των εξωτερικών χρηματοστικών ε, ροών για καλύτερη οικονομική διαφάνεια σε διεθνές επίπεδο. Συμφωνήσαμε με τη ΣΥΠΑ στον αφορά τον εντοπισμό των χρηματικών ροών, κυρίω των ροών εκείνων που χρηματοδοτούν στι δημοκρατικέ δράσει. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό επίση σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Τρίτη πτυχή, όταν αυτοί οι Ευρωπαίοι πολίτες εγκαταλείψουν την επικράτεια, πώς να χειριστούμε την επιτροπή τους στο ευρωπαϊκό έδαφος. Στις ευρωπαϊκές χώρες, όπως ξέρετε, υπάρχουν πολλές καλές πρακτικές. Έχουμε κάνει ακροάσεις και εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με αυτό και σχετικά με ένα δίκτυο που συλλέγει τις καλές πρακτικές. Νομίζω ότι αυτές οι καλές πρακτικές θα πρέπει να ενοποιηθούν και θα πρέπει να διαμορφωθούν σε μια στατικική ε, σφαιρική, διότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες ε, καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες ε, όσον αφορά την επιστροφή των πολιτών τους όταν επιστρέφουν στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Κάποιοι επιστρέφουν με συγκεκριμένο ε, αποφασισμένο τρόπο και μπαίνουν στο, πεδίο το ποινικό, άλλοι επιστρέφουν τρομοκρατημένοι, συγκλονισμένοι διότι είδαν και αυτούς τους νέους θα πρέπει να τους βάλουμε στις δέουσες δομές για να μην είναι πλέον ριζοσπαστικά στοιχεία. Κάποιες χώρες ε, αρχολούνται με αυτή την άπορη ριζοσπαστικοποίηση. Δεν θα πρέπει να μιλάμε συνέχεια γι' αυτό, αλλά κάθε μέρα βέβαια έχουμε επιστροφές ατόμων ε, που έχουν συγκλονιστεί ή έχουν υποστεί κάποια τραύματα ψυχολογικά και επιστρέφουν στο ευρωπαϊκό έδαφος. εξάλλου οι δικαστές που συναντήσαμε οι ίδιοι έχουν, ε, ε, δεν ξέρουν τι να κάνουν, λένε ότι τους έχουμε, τους ανακρίνουμε, τους ακούμε, τι κάνουμε μετά. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε εμεί, διότι η απάντηση θα πρέπει να δοθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα πρέπει να έχει πολιτική χρειά. Εν γέννη, αυτέ είναι οι γραμμέ τη εκθέσεω, οι βασικοί άξονε επί των οποίων επεξεργάστηκα τα συγκεκριμένα θέματα, εκεί που ακούσαμε στι ακροάσει διάφορε προσωπικότητε των ευρωπαϊκών χωρών. Λίγο πολύ, λοιπόν, αυτό είναι το υπόβαθρο και το σχέδιο τη εκθέσεω που σα υποβάλλω σήμερα και ευχαριστώ. Thank you very much, Σας ευχαριστούμε, κυρία Ντάτη. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και τόσο σύντομοι. Γιατί κατά το αναμενόμενο είναι μακρύτατος ο κατάλογος ε, των ομιλητών. Ε, με Ενδιαφέρει πολύ το ζήτημα πέραν αυτού. Ε, στις πολιτικές μας ομάδες έχουμε επεξεργαστεί πολύ το ζήτημα. Είναι πολύ επίκαιρο το θέμα. Θα ήθελα δύο πράγματα μόνο να πω υπογραμμίζοντας ε, όλα αυτά που έχουν γίνει για τους ε, ξένους αλλοδαπούς μαχητές και πώς ε, το δικαστικό μας σύστημα αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα της σπαστικοποίησης, στις φυλακές, το διαδίκτυο, όπως σωστά είπατε, γιατί αυτό το ζήτημα μας απασχολεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ξέρω ότι υπάρχει μια διάσταση απόψεων. Μπορεί να πω κάτι, δεν ξέρω αν θα οδηγήσει σε τροπολογίες ή θα γίνει μια ανταλλαγή απόψεων. Ε, ήθελα μόνο να μιλήσω για το θέμα της σύγκριση. Δηλαδή, είπατε για το Ηνωμένο Βασίλειο και ο κύριος Κύρκο που ξέρουμε ότι έχει μια σαφή τοποθέτηση για το ζήτημα. Υπάρχουν προγράμματα, ξέρω ότι παραδείγματος χάρη εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε σεμινάρια, και εγώ ε, ο ίδιος φέρνω ε, από τη χώρα μου ανθρώπους εδώ στο κοινοβούλιο. Όμως ε, αυτά που γίνονται αρκούν εκείνα και τα ποιοτικά στα κράτη-μέλη για τη σπαστικοποίηση. Παραδείγματος χάρη στις φυλακές γίνονται καλά πράγματα, καλές προσπάθειες. Στη δική μου τη χώρα Είχαμε ποιοτικέ προσπάθειες ε, σε περιφερειακή βάση, σε κάποιες φυλακές δηλαδή. Τι με απασχολεί όμως, ότι δεν είναι υψηλή ποιότητα αυτών των προγραμμάτων, ούτε και υπάρχει αντίστοιχη χρηματοδότηση. Αν γίνει μια σύγκριση ανάμεσα στις μεγάλες χώρες, τη Γαλλία, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, σε σχολεία, σε φυλακές, ε, τι ακριβώς συγκρίνεται. Και μετά, πέρα από τα, τη θρησκευτική διάσταση του ζητήματος, υπάρχει ε, η ψυχολογική πτυχή. Τώρα πλέον δεν μπορούμε να δίνουμε αφελείς ε, απλοϊκές απαντήσεις για, στο θέμα της ρησφοστικοποίησης. Ε, χρειαζόμαστε πραγματική ουσιαστική δράση. Για να δούμε. Η Άννα ε, είναι η πρώτη που ζήτησε τον λόγο. Ναι. Μάλιστα. Ξεκιν... Είσαστε σκιώδης, δεν είσαστε. Ναι, είμαι σκιώδης για την ομάδα μου. Και θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ρασίντα Ντάτσι για αυτό το έργο που αποτελεί πολύ καλή βάση για ε- την εργασία μας. Είναι πραγματικά περιεκτική και ευρεία Υπάρχουν τομείς που ακόμα και στη δική μου ομάδα κάποιοι μπορεί να διαφωνούν για κάποια διατύπωση. Την αναφορά, για παράδειγμα, για την ε, οδηγία διαβίβασης ε, προσωπικών δεδομένων των ταξιδιωτών, για παράδειγμα. Ωστόσο όμως από την άλλη πλευρά πιστεύω ότι είναι περιεκτικότατη αυτή η έκθεση, ευρύτατη και τα σχόλιά μου σχετικά και επίσης από την άλλη πλευρά πρέπει να πω ότι εκτιμώ το ότι δεν θέλετε να γίνεται λόγος για τα θρησκευτικά φαινόμενα ή θρησκευτικά αίτια που <clears throat> δεν ταυτοποιούνται ως τα κύρια στοιχεία σε αυτή την αντιπαράθεση και εκτιμώ την ευαισθησία σας και ευαισθητοποίησή σας σε σχέση με την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου με αυτόν τον τρόπο παρότι δεν θα μπορέσουμε να το αποφύγουμε να κάνουμε λόγο για την Ισλαμοφοβία πιστεύω διότι υπάρχει και αυτό το στοιχείο που αυξάνεται όλο και περισσότερο στην κοινωνία μας και είναι πολύ επικίνδυνο και δεν πρέπει να φοβόμαστε να το αντιμετωπίσουμε όμως κατανοώ τις ανησυχίες σας την ευαισθησία σας και τις εκτιμώ από την άλλη πλευρά τώρα πιστεύω επίσης ότι παρότι έχετε ένα κεφάλαιο σε σχέση με τους δεσμούς μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής ασφάλειας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ίσως θα μπορούσαμε ίσως να ήμασταν πιο εξειδικευμένοι, πιο συγκεκριμένοι και θα πρέπει βασιζόμενοι σε αυτά που μόλις μας αναφέρατε για την χρηματοδότηση της ε, τρομοκρατίας και τον ρόλο που διαδραματίζουν κάποιες χώρες χρηματοδοτώντας αυτή την ε, τρομοκρατία και δεν μπορούμε να αποφύγουμε το να μιλήσουμε για αυτό το πρόβλημα, τη Σαουδική Αραβία δηλαδή. Και κάποιοι σε σχέση με την Σαουδική Αραβία στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ΑΦΕΤ είχαμε τον Ευρωπαίο Συντονιστή κατά της τρομοκρατίας και όλο και περισσότερο πρέπει να έχουμε αυτή την ολοκληρωμένη προσέγγιση και πρέπει να έχουμε συναντήσεις της ΛΥΜΠΕ Πολιτικής Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και της ΑΦΕΤ Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων διότι αποτελεί πρόκληση για την εξωτερική μας πολιτική αυτό το φαινόμενο. Όμως σε αυτή τη συζήτηση εχθές κάποιος ανέφερε τη Σαουδική Αραβία σαν λέει μια μετριοπαθή χώρα. Λυπούμε που πρέπει να πω ότι εγώ εισηγήτρια για τη Σαουδική Αραβία και παρακολουθώ τις εξελίξεις εκεί, δεν είναι καθόλου μετριοπαθής χώρα. Και ιδιαίτερα όσον αφορά την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τα δίκτυα των δικτύων <clears throat> και σε σχέση με τη Σαουδική Αραβία που μπορεί να γίνεται στο τέλος τέλος και θύμα αυτών των τρομοκρατικών επιθέσεων είναι κάτι το οποίο όμως υφίσταται η εμπλοκή της Σαουδικής Αραβίας και δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε και να το αμελήσουμε και θα πρέπει να ε, συζητηθεί στο πλαίσιο της εκθεσής σας. Επίσης ε, ζητείτε να υπάρξει ένας κοινός ορισμός αλλοδαπών μαχητών, foreign fighters, αυτός ο ορισμός ε, αλλοδαπών μαχητών όπως υφίσταται σήμερα είναι κάτι απαράδεκτο. Είναι κατεφημισμόν ε, ε, ονομασία. Κάνουμε λόγο λοιπόν για τρομοκράτες, για εγκληματίες που πυκνώνουν τις γραμμές των τρομοκρατών και εμπλέκονται στις εχθροπραξίες. Οι άνθρωποι στο Ιράκ ρωτούσαν γιατί μιλάτε για αυτούς τους αλλοδαπούς μαχητές όταν είναι δικοί σας αλλοδαποί μαχητές είναι δικοί σας υπήκοοι αυτά τα άτομα γιατί να υιοθετούμε λοιπόν αυτήν την εφημιστική κατεφημισμό προσέγγιση ονοματίζοντας τους έτσι και να λέμε μαχητές ευρωπαϊκής προέλευσης ε, που εντάσσονται στις τρομοκρατικές οργανώσεις και δίκτυα και αποτελούν απειλή και πρέπει να σταματήσει ο προσιλητισμός και η κατήχηση ώστε να μην υπάρχουν όλο και νέοι νεόφοιτοι που κερδίζουν αυτά τα δίκτυα από αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει με σωστό τρόπο να εντάξουμε αυτό το θέμα ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί αποτελεσματική στι κοινέ δράσει των υπηρεσιών και οργανώσεών μα στο ευρωπαϊκό επίπεδο την τελευταία φορά που ε, επισκέφθηκα το κέντρο καταπολέμηση τη τρομοκρατία εδώ στι Βρυξέλλες μετά τι επιθέσει των Παρισίων, ξέρετε τι είδα. Είδα ότι δεν υπήρχε κανένα ειδικό ε, αραβομαθής, ε, ειδικό για τον αραβικό κόσμο και το Ισλάμ, που να παρακολουθεί από το διαδίκτυο και να επιβλέπει, να υποπτεύει το τι ε, τεκτενόταν. Είναι πραγματικά κεριότατα, κέρια στοιχεία αυτά και θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις οικογένειες όλες εκείνες που τα μέλη τους κινδυνεύουν ουσιαστικά και να κάνουμε πολύ καλύτερη δουλειά από πλευράς μας. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Συμφωνώ με την ευαισθησία που φαινόταν στο αρχικό κείμενο. Συνάδελφοι, είναι μακροσκελέστατος ο κατάλογος. Ξέρω ότι και εγώ δεν τήρησα τα δύο λεπτά. Αν μπορείτε να βοηθήσετε με δύο λεπτά ο καθένας κατά παρέμβαση, θα ήμουν ευγνώμων. Σκιώδης για το ECR, ο Τίμωθη Κίρκοπ. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο γρήγορος γίνεται. Σημαντικότατο θέμα. Το έχουμε εντοπίσει όλοι. Συγχαίρω την εισηγήτρια πρώτα απ' όλα. Πληρέστατη εισαγωγή. Συγκεκριμένες προτάσεις και προσεγγίσεις παρουσιάζονται. Θεωρώ ότι καλύπτουν τις προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση δυσχερέστατου προβλήματος. Θα ξεκινήσω βάσει ερωτήσεως. Τι είναι ρίζος παστικοποίηση. Το συζητούμε το λέμε και λέμε ριζοσπαστικοποίηση, ριζοσπαστικοποίηση, ριζοσπαστικοποίηση, από ριζοσπαστικοποίηση. Γιατί μιλάμε για κάποιους που κινούνται ριζοσπαστικά, δηλαδή εκτός των αποδεκτών ορίων της ε, σωστής περιφοράς, λόγω πολιτικής φιλοδοξίας, λόγω θρησκευτικών διαφορών, λόγω εξτρεμιστικών τοποθετήσεων κάποιων θρησκειών αυτό είναι δυσχεράστατο. Αν δείτε την κατάσταση εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, θα δείτε ότι η ρεσβαστική συμπεριφορά τώρα επί το παρόντο σε κάποιες χώρες της Μέσης Ανατολής τα διαπράττει τα χειρότερα, τα χειρότερα δικήματα διαπράττονται από, ε, από έναν κλάδο της θρησκείας έναντι άλλου κλάδου της θρησκείας. Οι Ευρωπαίοι πολίτες μας πηγαίνουν και πολεμούν για κάτι που πιστεύουν ότι είναι σοβαρός σκοπός. Συχνά, εάν επιβιώσουν και επιστρέψουν, επιστρέφουν απογοητευμένοι. Έχοντας όμως ριζοσπαστικές απόψεις και θέλουν να διαπράξουν αδικήματα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφερθήκατε στις ομάδες πριν. Είχα κάποια εμπειρία από αυτού. Εγώ αρνήθηκα όταν ήμουν στο Υπουργείο να μπουν κάποιοι άνθρωποι στη Βρετανία που είχαν κάποια συμπεριφορά τέτοιων θρησκευτικών ομάδων ε, και δοξασιών ε, που θα επηρέαζε πολύ ε, τους νέους και κυρίως θα ριζοσπαστικοποιούσε τη δεκαετία του 80 και 90 πολλούς νέους. Αυτό περιεκόπη και περιεκόπη το φαινόμενο λόγω παιδείας, εκπαιδεύσεως, αλλαγών, χρήσεως πόρων για να αποτρέψουμε τους νέους από το να ακολουθήσουν αυτή τη ριζοσπαστική προσήγγιση. Λοιπόν, πετύχαμε δηλαδή από ριζοσπαστικοποίηση. Λοιπόν, θέλω να πω εντάχει ότι ναι, θα πρέπει να περικόψουμε ε, τη χρηματοδοτής των ποινικών οργανώσεων, είτε είναι τρομοκρατικές οργανώσεις ή ποινικού δικαίου, να ανταλλάσσουν πληροφορίε μεταξύ κρατών με τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Είμαι απογοητευμένο. Υπάρχει έλλειψη ανταλλαγή πληροφοριών επικοδομητικών που μα χρειάζεται. Πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών. Η οδηγία για τα προσωπικά δεδομένα επιβατών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω θα βοηθήσει το Ευρωπαϊκό PNR. Τα εφιστάμενα μέτρα θα πρέπει να αναπτυχθούν έτσι περαιτέρω και νομίζω ότι σίγουρα ότι ποτέ δεν πρέπει να υποθέτουμε ότι για όλα αυτά το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο συμβάλλει στη ρίζοσπαστικοποίηση. Ακούσαμε ότι κάποιοι έφυγαν από τη Βρετανία να πάνε να πολεμήσουν και αφήσαν πίσω τους οικογένειες που ήθελαν την παστικοποίηση και θεώρησαν ότι τελικά ε, έπρεπε να υπάρξει αντιμετώπιση εντός της χώρας και ήταν πρόσωπο με πρόσωπο η ριζοσπαστικοποίηση. Και έτσι θα μπορεί να είναι και άπολη ριζοσπαστικοποίηση. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια έξοχη η εισαγωγή, έξοχη έκθεση και θέλουμε να την εξετάσουμε εκτενέστερα και περαιτέρω, αλλά είμαι ευγνώμων των εισηγήτρια για την πρωτοβουλία που ανέλαβε. Ευχαριστώ Τιμόθη. Νομίζω ότι πολλοί από, απ' έξω θα διαβάσουν την έκθεση, θα εξετάσουν τα θέματά της. Μπορεί να έχουμε πρόβλημα αν μακρηγορούμε, ένα πρόβλημα είναι ότι δεν θα μπορούμε να εξετάσουμε τη δική μου έκθεση που ακολουθεί. Δεν το βλέπετε σαν πρόβλημα πιθανώς εσείς. Τέλος πάντων. Καλώς. Σκιώδης της Μάιτε. Ναι, θα προσπαθήσω να περιοριστώ σε αυτά τα δύο λεπτά και να μην τα ξεπεράσω. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσουμε την εισηγήτρια για τη δέσμευση και την προσπάθεια. Είναι αξιοπρόσεκτη η προσπάθεια που έκανε και προσπάθησε ακριβώ να ανταποκριθεί σε αυτό το οποίο ζητεί και η Επιτροπή. Μια συνολική σφαιρική στρατηγική. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε, δεχόμενοι όλα τα σημεία που, ε, πρέπει, που εντάσσονται στην έκθεση, να αλλάξουμε του ανθρώπου σε σχέση με την σύλληψη, κράτηση, ε, καταστολή σε σχέση με τους Ευρωπαίους πολίτες. Ή θα προσθέσουμε την ε, καταστολή ή θα αφαιρέσουμε άλλα εδάφη. Εκείνο το οποίο κάνουμε είναι να στείλουμε ένα μήνυμα πολύ σαφές προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό που θα πούμε είναι ότι η δική μας άποψη για τη δράση μας είναι ότι στη στρατηγική κατά της τρομοκρατίας και την υπεράσπιση της δημοκρατίας πρέπει να είμαστε σφαιρικοί σε ολοκληρωμένο πλαίσιο. Αν το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι πρόληψη σε σχέση με τη ριζοσπαστικοποίηση, υπάρχουν και άλλα πράγματα Διαφορετικά πρέπει να προσθεθεί και το θέμα της καταστολής ε, για να, είμαστε, να συνάδει ο τίτλος με την ουσία του περιεχομένου. Πρέπει να είμαστε συνεκτικοί μεταξύ του τίτλου και του περιεχομένου. Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε είναι σαφέστατο. Είτε είναι ο ένας είτε ο άλλος ο τίτλος αυτής της έκθεσης. Ζητούμε μια σφαιρική στρατηγική, διότι μόνο σφαιρικά ολοκληρωμένα θα μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε ή να, ε, ε, α, να σβήσουμε, να εξοντώσουμε αυτό το φαινόμενο της τρομοκρατίας. Λοιπόν, ολοκλήρωση. Σε σχέση με την κοινωνία, ολοκλήρωση και ένταξη αυτών των πιο ευάλωτων στοιχείων που κινδυνεύουν να ριζοσπαστικοποιηθούν και να αποκλειστούν. Άλλο μήνυμα και θα προσπαθήσω να περιοριστώ στα δύο λεπτά και να μην τα ξεπεράσω για να ενισχύσουμε, να ενδυναμώσουμε το τμήμα εκείνο που εμείς ακόμα δεν έχουμε αναπτύξει επαρκώς και που είναι η πρόληψη και η απορριζοσπαστικοποίηση, ραν, το δίκτυο αυτό κατά της, για την ευαισθητοποίηση για τη ε, ριζοσπαστικοποίηση πρέπει να έχει διαφορετικό περιεχόμενο από το σημερινό το RAN, το δίκτυο ευαισθητοποίησης για την ε, ριζοσπαστικοποίηση, έχει περιορισμένα κονδύλια, έχει μια στρατηγική που ακόμα μόνο θέτει σε επαφή κάποιες καλές πρακτικές ε, ως απόθεμα, αλλά δεν υπάρχει ούτε η εκμετάλλευση του ενός στο ένα δέκατο όλων αυτών των δυνατοτήτων. Η έκθεση δεν είναι, ε, που αφορά αυτά δεν είναι το πιο σημαντικό τμήμα λοιπόν σε σχέση με αυτά. Πρέπει με ρητό τρόπο να αναφερθούμε στην πρόληψη και από ριζοσπαστικοποίηση ή να αναπτύξουμε περισσότερο αυτό το τμήμα ή να στείλουμε το μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι και να πούμε ακόμα βρίσκονται στα σπάργανα αυτού του είδους ε, οι δυνατότητες. Πρέπει να προχωρήσουμε πολύ πιο πέρα στη φαρέτρα και στον εξοπλισμό ε, από τις βέλτιστες πρακτικές Πρέπει να ενδυναμώσουμε με ειδικό ε, έκτακτο τρόπο αυτές τις δυνατότητες αυτές τις οποίες ε, είδε και ε, παρίτμησε η κυρία Ρασίντας ε, Ντατή πρέπει να γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα να μπορέσουν να ευδοκιμήσουν και πώς μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα τα πράγματα οι ανταλλαγές αστυνομικών αρχών και οι βέλτιστες πρακτικές κτλ. Και μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Σε σχέση με το ειδικό τμήμα για την ζωσπαστικοποίηση πρέπει να το αναπτύξουμε περισσότερο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ η Μπάρβαρα Σπινέ. Δύο ή τρία λεπτά. Μπάρμπαρα, όλοι θέλουν, ε, μιλούν περισσότερο από την κυρία Τάτη. Κοιτάξτε συνάδελφοι, κοιτάξτε, έχει μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό θέμα. Και υπάρχει μεγάλη εμπειρία ενδιαφέρον, δεν κατηγορώ τους συναδέλφους που μακρηγορούν. Α δυστυχώς έχουμε και ψηφοφορία βλέπετε. Παρακαλώ. Πειθαρχία παρακαλώ. Και έχουμε και τροπολογίες που θα υποβάλουμε και μπορούμε να το εξεργαστούμε. Ακολουθήστε την κυρία Ντατή, σαν παράδειγμα, που ήταν συντομότατη στην εισαγωγή που έκανε. Πάνω απ' όλα θα ήθελα να πω ευχαριστώ στη Ρασίν Ντατή για την έκθεσή τη, Τη μελέτησα ευρέω για το θέμα της απόρριζας Κάποια σημαντικά θέματα υπογραμμίζει, είναι οι βασικές επαφές με τα θύματα, η αναγνώριση του έργου των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των διαφόρων φορέων της κοινωνίας των πολιτών και για το συμπέρασμα όσον αφορά την ε, πρόληψη και καταστολή. Αλλά εδώ αναφύονται κάποιες αμφιβολίες για μένα και κάποιες βελτιωτικές προτάσεις μου. Η αμφιβολία αφορά την τοποθέτηση τη γενική που είναι αντιβαίνει θα έλεγα τον τίτλο. Δηλαδή την αρχική πρόταση όσον αφορά την πρόληψη σε σχέση με την καταστολή. Νομίζω ότι ενοποιούνται τα δύο πράγματα και στο τέλος καταλήγουμε σε προληπτική καταστολή. Ελαφρώς ανησυχητικό που θυμίζει και την ταινία Minority Report. Τώρα θα σε κάποια στοιχεία. Πρώτο, η ριζοσπαστικοποίηση στις φυλακές. Έχω κάποιες αμφιβολίες όσον αφορά της απομόνωσης εντός ε, των φυλακών. Γκέτο μέσα στο γκέτο. Είναι μια εμπειρία που τη γνωρίζω πολύ καλά στην Ιταλία. Εφαρμόζεται στους μαφιόζους, στους πιο επικίνδυνους. Και δεν ξέρω αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην απορριζοσπαστικοποίηση δηλαδή και έναν ενδεχόμενο τρομοκράτη, δυνάμει τρομοκράτη που δεν έχει ακόμα διαπράξει δικήματα. Μετά είναι η πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης στο διαδίκτυο. Έχω ανησυχίες σχετικά με αυτό. Θεωρώ ότι ο έλεγχος του διαδικτύου πάντα είναι κάτι ακαθόδες. Ε, υπενθυμίζω ότι εσείς ορίζετε το διαδίκτυο σαν εικονικό πεδίο για τους δυσπροσφαστικούς τρομοκράτες. Μου υπενθυμίζει αυτή η φράση κάτι που είπε πριν από μερικές μέρες ο Ομπέρτο Έκο, συγγραφέας το διαδίκτυο, είναι το εικονικό πεδίο των ανοήτων. Είναι δύο ε, θέσεις που δεν μπορώ να δεχτώ. Κάτι άλλο που αφορά την εκπαίδευση και την ένταξη. Θεωρώ ότι είναι θεμελιώδου σημασία, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε όσον αφορά τη μουσουλμανική θρησκεία. Πιστεύω ότι χρειάζεται πραγματική κατάρτιση και εκπαίδευση των ημάμιδων ε, και η πρόθεση του το έργου τους στις φυλακές και τέλος το PNR, τα προσωπικά στοιχεία των επιβατών. Εγώ και η ομάδα μου είμαστε εναντίον Ε, της θέσπισης αυτού του μέτρου. Κλείνω. Τέλος, η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις χώρες του κόλπου όσον αφορά τις οικονομικές ροές. Συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι κάτι. Να θυμηθούμε ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών έχει αποτύχει κτρά. Η συνεργασία με τις χώρες του κόλπου θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά παρακινδυνευμένη βλέποντας τη χρηματοδότηση που χορηγούν στο Ισλαμικό κράτος. Υπενθυμίζω επί ευκαιρία του Ισλαμικού κράτους ότι χρηματοδοτήθηκε αρχικά και από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Χρηματοδοτούσαν, είπα, και το Ισλαμικό κράτος στην αρχή. Ευχαριστώ πολύ, Μπάρμπαρα. Το πέρασε όλα τα μηνύματα. Ευχαριστώ. Και η Τζιν, η για τους Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για αυτή την έκθεση που μας ε, που εμπεριέχει πολλά σημαντικά στοιχεία όπως το έτσι Παραδείγματο χάρη σε σχέση με το, τη διάσταση των πολιτικών ελευθεριών και των ατομικών δικαιωμάτων. Ε, έχω θέμα με τον ορισμό όπως και ο Τίμωθη. Ακριβώς νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε το τι εστί ριζοσπαστικοποίηση. Πρέπει να, να δούμε πώς ακριβώς προκύπτει η σύνδεση με τις ριζοσπαστικές πολιτικές ιδέες. Τώρα, ε, όταν μιλάμε για το τι συμβαίνει στην Ουκρανία στα σύνορα με τη Ρωσία, ε, μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν και Ευρωπαίοι μαχητές. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για αντιπαλώτες ανάμεσα σε παρακλάδια μίας ε, και μόνο θρησκευτική ιδεολογίας. Ε, και σε σχέση επίσης με την παστικοποίηση θα πρέπει να δούμε πώς ακριβώς ε, θα αντιμετωπίσουμε και υποψίες ε, για μέλη των δικών μας κοινοτήτων. Τώρα, ε, το άλλο ζήτημα είναι το κράτος δικαίου με τις συζητήσεις που έχουμε κάνει στο Κοινοβούλιο για τη σχετική νομοθεσία για την παρακολούθηση στο ίντερνετ, την ασφάλεια στο ίντερνετ και ούτω καθεξής. Στο κομμάτι για την παιδεία επίσης ε, υπάρχει το θέμα της ενσωμάτωσης και της κριτικής σκέψης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ως προς την πρόληψη που επιχειρούμε να προωθήσουμε για να καταπολεμήσουμε την ριζοσπαστικοποίηση. Ε, για τα στοιχεία επιβατών, το PNR, νομίζω ότι αυτό δεν σχετίζεται απαραίτητα με την πρόληψη της άπορης Και νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να μας απασχολήσει σε συνδυασμό με τον ορισμό, δηλαδή η γεωγραφική συνιστόσα. Κάποιος που πάει στο κουμπάνι και υποστηρίζει τους Κούρδους και κάποιος που θα ε, αγωνιστεί στο πλευρό του Ισλαμικού στρατού είναι ένα και το αυτό. Αυτό θέλω να το ξέρω. Τι εννοούμε ακριβώς. Για την επιστροφή των μαχητών πρέπει να συνοηθούμε. Επίσης, ε, ε, δεν μπορούμε για τις γλώσσες να περιοριστούμε στα αραβικά, στο Ουγγντού παραδείγματος χάρη. Δεν έχουμε ε, πραγματογνωμοσύνη. Αφήστε που υπάρχει και το ζήτημα των δύο φύλων και κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε γι' αυτό. Πάντως, πολύ καλή αρχή. Ναι, Τζιν, ευχαριστούμε. Κριστίν, ε, ε, από την DG Home. Ε, ευχαριστώ την Ρασίδα Τατή, κάνει διάφορες διαπιστώσεις, παρατηρήσεις και μας δίνει ιδέες για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης. Τονίζεται η προσθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και τη στρατολόγηση των αλλαπών μαχητών. Όμως θα πρέπει να τονίσουμε και κάποιες επιτυχίες της ριζοσπαστικοποίησης που δεν αναπτύσσονται μέσα στο σχέδιο έκθεσης και θα καταθέσω τροπολογία τροπολογίες σχετικές. Οι ρίζες ε, της ρίζοσπαστικοποίησης ε, δεν, ε, μας δεν μπορούμε ίσως να αντιληφθούμε το εύρος του φαινομένου, αλλά να δείξουμε τουλάχιστον δεν υπάρχει ομοιομορφία και να τονίσουμε ότι οι παστικοποιημένη ή ή οι ρίζος ε, δεν οθούνται μόνο από τη θρησκεία. Αυτό είναι μόνο ένα κίνητρο, ένα παράγοντας. Πέραν αυτού, ε, το διαδίκτυο ε, μπορεί να αναδειχθεί και σε πλατφόρμα αντιλόγου σε σχέση με την στρατολόγηση ε, και την προσπαστικοποίηση και να προωθεί τις αξίες μας της ανεξιθρησκείας, της συμβίωσης, της ελευθερίας έκφρασης. Επίσης, πέρα από την πάταξη της ριζοσπαστικοποίησης και την καταπολέμηση των τρομοκρατικών δράσεων αυτών των ριζοσπαστικοποιημένων θα πρέπει να βοηθήσουμε και να προωθήσουμε την ενσωμάτωσή του στην κοινωνία αποριζοσπαστικοποιώντας έτσι την, ε, την ίδια την κοινωνία και αυτές τις κοινότητες και το, προωθώντας την αυτονομία επίσης των νέων. Ε, δεν θα πρέπει μόνο να καταδικάζουμε απλές ιδέες αλλά την προσφυγή στην βία που είναι κάτι απαράδειγμα έκρηκτος. Σας ευχαριστούμε, Κριστίνε. Ήσασταν συνοπτικότατοι. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ ενώνω τη φωνή μου με τους προλαλήσαντες ε, που επένεσαν το έργο της κυρίας Ντατή. Δεν θα προσθέσω τίποτα, διότι πιστεύω ότι ήδη υπόθηκαν πολλά καλά λόγια. Κάποια σχόλια. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι στην έκθεσή της η κυρία Ντατή είναι λίγο αυστηρή όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επίτροπη, κυρίως όταν ζητά το συντομότατο να καταστεί σφαιρική ε, στρατηγική που θα αποφύγει θατολόγηση και θα οδηγήσει στην απορριζοσφαστικοποίηση. Ε, είχα διαβάσει κάτι το 2014 που αφορούσε αυτό το στόχο, σχετικό κείμενο. Υπάρχει ένα στοιχείο επικαιροποίηση που απαιτείται, που θα πρέπει να λάβει η χώρα. Ε, έχω κάποια στοιχεία που θεωρώ ότι θα πρέπει να ενημερωθούν δεν μιλάμε για την μονάδα που θα λειτουργήσει εντός της Ευρωπόλ την 1η ε, Ιουλίου ε, που πρέπει να δημιουργηθεί. Πρέπει να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία, τα σπονή, τη μονάδα που θα είναι αρμόδια για την ε, ανοχή κλπ. Όσον αφορά για τις δυνατότητες που υπάρχουν σε κεντρικό επίπεδο και τις εθνικές δυνατότητες, όσον αφορά το διαδίκτυο. Λέτε ότι κάθε κάτω μέλος θα έπρεπε να δημιουργήσει μια μονάδα ειδική που θα ασχολείται με το διαδίκτυο και το παράνομο περιεχόμενο. Είμαι πεπισμένο ότι θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα επιχειρησιακά αν μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα αυτά σε επίπεδο τη Ευρωπόλ. Και νομίζω ότι αυτή είναι η αποστολή τη Ευρωπόλ και να δημιουργήσουμε τι συνθήκε όπου να μπορούν να υλοποιηθούν αυτά. Διότι μπορούμε να ακολουθήσουμε την ορμή αν υπάρχει μια ομάδα ε, και βλέπουμε τι θα γίνει σε μια, στην Ελβετία, στη, στο Λουξεμβούργο, στη Γερμανία, στην Αυστρία ε, να ασχολείται κάθε ομάδα και να συλλέγει τα στοιχεία. Για το περιεχόμενο το παράνομο, οι πάροχοι του διαδικτύου αντιδρούν πάρα πολύ γρήγορα όταν υπάρχει η Ευρωπόλ που κινεί το όνομα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω που του ζητεί να αποσύρουν επικίνδυνο περιεχόμενο παρά μια μικρή χώρα που απευθύνεται προ του παρόχου. Εκεί νομίζω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που θα πρέπει να διευκρινιστούν. Ε, τώρα, υπάρχουν κάποια σημεία που θα είναι πάρα πολύ ευαίσθητα και νομίζω ότι θα πρέπει να επανεξετάσουμε τη διατύπωση. Το σημείο 9, όταν μιλάτε για ποινικέ κυρώσει, θεωρώ ότι η διατύπωση δεν είναι επαρκή. Ποινικέ κυρώσει δεν μπορούν να απευθύνονται για κάποιον που δεν αντιδρά. Οι ποινικέ κυρώσει απευθύνονται προ κάποιον που κάνει κάτι το οποίο δεν είναι ορθόν. Υπάρχουν στοιχεία τα νομικά που πρέπει να διορθωθούν. Και στο σημείο 21 για το PNR. Θα σταματήσω με δύο σκέψεις. Θεωρώ ότι υπάρχει κάτι εκτός της εκθέσεως που θα πρέπει να έχουμε επίγνωση αυτού και το συζητήσουμε. Ε, λοιπόν, υπάρχουν, δεν φεύγει οποιοδήποτε να πολεμήσει επηρεάζονται από το περιβάλλον τους αυτοί που πάνε να πολεμήσουν. Η καταπολέμηση της λαμοφοβίας ε, και της απομόνωσης είναι προαπαιτούμενο για την άπορη ζωσπαστικοποίηση και την καταπολέμηση της ζωσπαστικοποίησης. Εκείνοι που θέλουν να φύγουν θέλουν να ζήσουν μια εποπία ε, και θέλουν να νικήσουν. Άρα στόχος θα πρέπει να είναι δημιουργηθούν οι συνθήκες τις οποίες η ΝΤΑΕΣ θα συνθλιβεί στατιωτικά. Δεν θα πάνε σε σταυροφορία κάποιοι αν δεν ε, θέλουν τουλάχιστον, αν δεν έχει ε, τουλάχιστον κερδιθεί μία μάχη. Άρα δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η δόξα και οι νίκες. Ο Τόμας είναι επόμενος που έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κλοντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή την έκθεση ε όχι την παρακολούθησα και θέλω κάποιες σύντομες παρατηρήσεις να κάνω. Χαιρετίζω αυτή την έκθεση ως μια ευρεία περιεκτική πλήρη έκθεση που είναι μια καλή απεικόνηση των γεγονότων και στοιχείων αντικειμενικά. Το χαιρετίζω, την χαιρετίζω στην έκθεση. Ο ρόλος των σχολείων και των συστημάτων παιδείας και εκπαίδευσης που τονίζει η συγγήτρια είναι κάτι που υποστηρίζω και εγώ. Αλλά επίσης και η κοινωνία και οι κοινότητες και η οικογένεια διαδραματίζουν ρόλο, οι οικογένειες ε, και όχι μόνο τα σχολεία. Για παράδειγμα, λέσχες ελεύθερου χρόνου που ακολουθούν για την απασχόληση τέλο πάντων την παρακολούθηση κάποιων πραγμάτων από τα παιδιά μετά το σχολείο διαδραματίζουν ρόλο και αυτές οι λέσχες πρέπει να μάθει κανείς από παιδί να μαθαίνει κανείς από παιδί τους πιο αδύναμους πρέπει να προστατεύουμε και να μαθαίνουν οι νέοι αυτές τις αρχές και να εξοικειώνονται με αυτές. Ένα τελευταίο στοιχείο που θέλω να αναφέρω εδώ είναι το εξή. Με ικανοποίηση παρατηρώ ότι η κυρία Ντατή δεν φοβάται να κάνει λόγο εδώ και για τα πιενά, τα προσωπικά δεδομένα ταξιδιωτών και τη διαβίβασή τους. Διότι πιστεύω ότι το PNR είναι ένα πολύ σημαντικό συστατικό στοιχείο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και θέλω σίγουρα να επενέσω το θάρρος της ε, για το ότι ανέφερε αυτό το... Thank you very much. Η Βρυγίτη ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και ταυτόχρονα θα ήθελα να ρωτήσω ακριβώς γιατί πράγμα μιλάμε, διότι διαβάσατε την έκθεσή σας μπερδεύτηκα. Κάνουμε έκθεση για την αντιτρομοκρατική δράση ή για την πρόληψη της ρίζος παστικοποίησης. Αλληλένδετα μεν τα ζητήματα, διαφορετικά δε. Το PNR είναι θέμα αντιτρομοκρατίας και όχι πρόληψης της ε, ριζοσπαστικοποίησης. Θα ήθελα λοιπόν να είναι, παραμείνουν διακριτά τα ζητήματα και να ε, συντάξετε μια έκθεση για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης γιατί για την αντιτρομοκρατία έχουμε έκθεση μάλλον για την καταπολέμηση της για την κατάσταση στις ε, φυλακές. Όντως, πρόκειται για φυτόρια ριζοσπαστικοποίησης. Όμως, τι θα θέλετε να κάνουμε, να θέλουμε στις φυλακές ε, τους καλύτερους ημάμιδες. Ε, ε, ξέρετε τι, ποιο είναι το πρόβλημα, ε, ότι τα σοφρονιστικά ιδρύματα είναι υπερφορτωμένα και ότι δεν έχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες οι φύλακες. Και ε, υπάρχουν κάποιοι που ακούνε κάποιες ε, ιδέες και τους υπόσχονται, οι μάμοι τους υπόσχονται μεγαλύτερη ζωή όταν ε, φεύγουν από τις φυλακές, αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Ε, για το διαδίκτυο. Είπατε ότι επίσης είναι αιστεία ριζοσπαστικοποίηση. Συμβαίνει αυτό όμως, θα συμφωνήσω με τον Τίμο Κύρκοπε. Το διαδίκτυο είναι ένα εργαλείο που μη δίνει ε, και καλή και κακή καθοδήγηση. Λοιπόν, η κακή καθοδήγηση είναι για την ρίζοσπαστικοποίηση. Μας οδηγεί στην ρίζοσπαστικοποίηση. Ε, όμως ε, πρέπει να καταλάβουμε ότι το εργαλείο από μόνο του δεν αρκεί. Υπάρχει κάποιος από πίσω, ένας άνθρωπος από πίσω που ε, σας καθοδηγεί, που μπορεί να σας ε, βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε σωστά το ίντερνετ, να ξέρετε τι ψάχνετε. Για τα καρτούν τώρα, τα που γεννούν τη βία. Συγγνώμη, αλλά κανένα εικονογραφημένο δεν μπορεί να γεννήσει βία. Η πολιτική ομάδα που καταχράτε, τα καταχράτευε υπέρ τη ιδεολογίας του για να ενισχύσει την εξουσία του, ε, οδηγεί μετά από παραπλάνηση σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή τη βία. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ε, αυτολογοκρισία. Α, μήπως αυτό είναι υπέρ τη στάδια της δύναμη τρομοκρατικής ομάδας μα είμαστε, ζούμε σε ελεύθερη ήπειρο δεν μπορούμε λοιπόν να περιορίζουμε εμείς ε, τις ελευθερίες μας και να αυτολογοκρινόμαστε θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τις ε, ε βασίτερες ε, τις ε, πραγματικές ρίζες της ρίζοσπαστικοποίησης και να μην κρυβόμαστε τη, μία από τις απαντήσεις θα τις βρούμε στις δικές μας εγχώριε πολιτικές σας ευχαριστούμε ε, Μπεργίτε ή Μαριών. Ευχαριστώ. Απηχώντας αυτά που είπε και η Μπίργκιτ, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά που είπε και ο Τίμωθη, είναι προφανές ότι α, οξύνει ε, τάσεις, ε, υφέρπουσες τάσεις κοινωνίας το διαδίκτυο και ελοχεύει ο κίνδυνος μέσω της καταστολής του διαδικτύου να ε, οξύνουμε ε, με αυτή τη δράση την ε, βία, την ριζοσπαστικοποίηση. Ε, την περαιτέρω, γιατί ξέρετε είναι και ευαίσθητο λεπτό το ζήτημα και υπάρχουν μεγάλα πάθια από τις δύο πλευρές. το διαδίκτυο δεν είναι ε, πλατφόρμα για ε, λογοκρισία. Το αντίθετο σημαίνει το ίντερνετ. Χρειαζόμαστε μια δικαστική απόφαση για το παράνομο περιεχόμενο. Δεν μπορεί απλώ επειδή ισχυρίστηκε κάποιο ότι πρόκειται για παράνομο περιεχόμενο να ανακηρυχθεί σε παράνομο περιεχόμενο. Δύο πράγματα χρειαζόμαστε λοιπόν παρακολούθηση από πλευρά των αστυνομικών δυνάμεων ή των αρχών επιβολή του νόμου ε, και, εν πάση περιπτώσει, με κάποιο ένδικο μέσο να κρυθεί ε, το περιεχόμενο διότι παρακινεί σε μίσωση, σε πράξη, σε βία. Αυτό είναι ένα πράγμα. Άλλο πράγμα είναι ε, η κοινωνική παρακολούθηση, όπω λέγεται, social monitoring και αυτό γίνεται από τι οργανώσει κοινωνία των πολιτών, από τι μη κυβερνητικέ οργανώσει ε, και εκεί πέρα ε, πρέπει να αναπτύξουμε τον αντίλογο, όχι από ειδικού σε προπαγάνδα, αλλά με κάποιου που θα είναι η δουλειά του αυτό, θα ασχολούνται με αυτό. Και όντω τέτοιε δράσει ε, θα πρέπει να τι στηρίξουμε. Όμω εκεί εντοπίζω ελλείψη, εκεί χωλαίνει η πολιτική μα. Σα ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρο. Ε, αναφέρθηκαν πολύ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, πρωτού περάσουμε στο πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα και εγώ ε, και κλείνοντας έτσι και τον κατάλογο των μιλητών να, να κάνω μια ερώτηση. Μιλάτε στο κεφάλαιο 7 για την ριζοσπαστικοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών. Νομίζω η Ντίν Λάμπερ και ο Τίμωθη Κύρκο που θα συμφωνήσουν ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και όχι μόνο στο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο κύριος Ντιπρέ αναφέρθηκε σε αυτό, ένα, μια αιτία επαναριζοσπαστικοποίηση ε, είναι ε, όταν, με, άμα την επιστροφή των ε, ανθρώπων αυτών και λόγω των προβλημάτων στο ασφαλιστικό σύστημα ή στο σύστημα περίθαλψης υγείας επαναριζοσπαστικοποιούνται. Λοιπόν, θεωρείται ότι είναι σοβαρό αυτό το ζήτημα και πρέπει να ασχοληθείτε με, στην έκθεσή σας και να τονίσετε αυτό το σημείο, διότι ξεκάθαρα είναι εθνική αρμοδιότητα, όμως είναι ε, ε, σοβαρή αιτία ρίζος όμως θα έπρεπε να το πραγματευτείτε και αυτό. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα τον Υπουργό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά, κυρία Ντάτη, θα σας ακούσουμε σας για να απαντήσετε. Ένα λεπτάκι, το συνάδελφο ρωτάω ζητήσατε το λόγο. Συγγνώμη, αλλά εγώ δεν σας είχα καταγεγραμμένο εδώ στον κατάλογο. Λοιπόν, Επιτροπή Κυρασίντα στο, στο τέλος. Ολιβιέ. Thank you, Chair, and thank you for... Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ που μας προσκαλέσατε σήμερα εδώ. Πραγματικό, πιστεύω πραγματικά ότι η τακτική ανταλλαγή απόψεων μπορεί να βελτιώσει την κατανόηση και τη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων μα. Ευχαριστώ λοιπόν. Σημαντική έκθεση αυτή. Ένα θέμα σημαντικό που φτάνει σε κατάλληλη στιγμή. Σημαντική όχι μετά τα γεγονότα τη Τίνιδα και των Παρισίων κλπ. Διότι τη στιγμή που συζητούμε, οι Υπουργοί Εσωτερικών συζητούν συζητούν το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ασφαλείας που πρότεινε 27 Απριλίου που πέρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πράγματι λοιπόν Κάποιες πρωτοβουλίες και προτάσεις ήδη έχουν διατυπωθεί και δράσεις έχουν δρομολογηθεί επιγραμματικά και τηλεγραφικά. Συμμεριζόμαστε την άποψη ότι η ριζοσφαστικοποίηση είναι περίπλοκος, περίπλοκη διαδικασία και από ριζοσφαστικοποίηση που δεν είναι ε, μονοπόλιο φιλοσοφία, πίστης ή πολιτικού συστήματος. Οι εκθέσει της Ευρωπόλη είναι σαφέστατες, Υπάρχουν πέντε μεγάλες πηγές και κίνητρα, αν θέλετε, που κινητοποιούν τη ριζοσφαστικοποίηση. Η θρησκεία είναι μία από τις αιτίες. Θα πρέπει να μη στιγματίζουμε λοιπόν. Δεύτερον, η θρησκεία αυτή αυτή, κατά την άποψή μας, δεν είναι το βαθύ αίτιο, το βαθύτερο αίτιο, αλλά η κατάχρηση αυτής. Ή θα έλεγα οι απλουστευμένες ερμηνείες από κάποιους της θρησκείας και σε παγκοσμιοποιημένο κόσμο, σε κάποιους που πάσχουν αποστές και ε, αβεβαιότητα, ε, είναι εύκολα θύματα. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε, πώς να πω, να το πω μια ανάλυση ε, με αποχρώσεις όσον αφορά τα αίτια. Θα πρέπει όμως την απάντηση να είμαστε στεναροί και άτεγκτοι. Τώρα όσον αφορά την πρόληψη, όπως λέμε στα γαλλικά, το soft is the hardest. Λοιπόν, μιλάμε για εκπαίδευση, για ενσωμάτωση, σοφρονιστικά συστήματα, καλές πρακτικές, επαφές με τους first liners δηλαδή με αυτού που είναι επιτόπου, όλα αυτά δεν παράγουν αποτελέσματα μια νυχτή. Είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε. Θέλουμε να δώσουμε απαντήσει με αποχρώσει ώστε σε ένα περίπλοκο πρόβλημα, ε, όντε ταχύ και αποτελεσματική. Υπάρχει αντίφαση ε, που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι Υπουργοί. Από πλευρά πολιτική βλέπω ποια είναι η πρόκληση λοιπόν. Ναι, έχουμε εμεί προτείνει μια τροπολογία όσον αφορά την απόφαση πλαίσιο που καθορίζει την τρομοκρατία για να συμπεριλάβουμε και το φαινόμενο των ξένων μαχητών συμπελαβανομένου και το άλλο γεγονότος ότι εκπαιδεύονται στο εξωτερικό αυτοί. Έχουμε διατυπώσει και κάποιες προτάσεις πολιτική ε, πολιτικής, η τελευταία είναι 28 Απριλίου, για τη ριζοσφαστικοποίηση πέρσι, ένα σχέδιο δράση με 16 σημεία ε, που εξετάστηκε από το, το Δεκέμβριο του Συμβούλιο επ' αυτού. Εγώ μπορώ να συζητήσω τα διάφορα θέματα λεπτομερώς άμα θέλετε, αλλά όσον αφορά τι καλέ πρακτικέ και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ευαισθητοποίηση για τη ριζοσπαστικοποίηση, το ράν. Ε, ακούσαμε το μήνυμά σας. Ε, από το μήνα Σεπτέμβριο ο προπολογισμό του δικτύου ε, θα πενταπλασιαστεί. Από 20 άτομα που είχαμε εδώ και 4 χρόνια έχουμε πάνω από 1.500 οργανώσεις. Δεν μιλώ για άτομα, μιλώ για 1.500 ενώσεις, ομοσπονδίες, πλατφόρμες, μη κυβερνητικές οργανώσεις που ε, ημερησίως εργάζονται, είτε είναι αστυνομικοί, είναι οι λέσχες, οργανώσεις νεολαίας κλπ, σοφρονιστικοί υπάλληλοι, ε, οι οποίοι εργάζονται καθημερινά για την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Αλλά όχι μόνο αυτό. Δεν πρόκειται απλώς ε, περί να, υπάρχει ένας κατάλληλος καλών πρακτικών ε, online. Περάσαμε σε ένα στάδιο που τώρα προσφέρουν μια υποστήριξη, συμβουλές κατόπιν αιτήματο σε κάποια τα κράτη-μέλη. Αυτή λοιπόν η λειτουργία θα ενισχυθεί από το μήνα Σεπτέμβριο. Δηλαδή μια στήριξη που απηχεί τι απόψει των ειδικών, εκφράζει την άποψή του που στρέφεται προ πολιτικού. Κάθε 18 μήνες, ένα χρόνο στους δύο, οργανώνουμε μια διπυργική διάσκεψη όπου καλούμε και εκείνους που ασχολούνται στην πράξη με το δίκτυο και τους υπουργούς εσωτερικών να ανταλλάσσουν απόψει. Και τολμώ να πω, γίνεται και μια αντιπαράθεση ιδεών. Τι λείπει, τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί, τι γίνεται σε εθνικό επίπεδο, τι πρέπει να γίνει σε εθνικό επίπεδο, τι πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλα αυτά τα μηνύματα λοιπόν ε, έχουν εισακουστεί Όσον αφορά το διαδίκτυο, πράγματι, πράγματι τη μεγάλη πρόκληση είναι να διατηρήσουμε την ελευθερία αυτό του φανταστικού εργαλείου που είναι το διαδίκτυο, αποφεύγοντας ε, περιεχόμενο να υπάρχει που δεν δεχόμαστε στο περιοδικό. Το Inspire της al δεν θα δεχόμαστε σε χάρτινη έκδοση να πωλείται. Γιατί να είναι διαθέσιμο ε, στο διαδίκτυο. Λοιπόν, η προσέγγιση που ακολουθήσαμε είναι να συμμετάσχουν οι φορείς του τομέα. Δημιουργήσαμε μια πλατφόρμα, είμαι σε επαφή ε, με αυτού ζητούν να εξηγήσουν τι κάνουν, ποιοι είναι αυτοί. Και υπάρχει νομική πτυχή, ε, υπάρχουν περιεχόμενα που είναι σαφώ παράνομα, ε, υπάρχουν περιεχόμενα που είναι ριζοσπαστικά, αλλά τον έχει κανείς ακραίε σκέψει και ακραίες απόψεις στις δημοκρατικές κοινωνίε δεν είναι αδίκημα. Το θέμα είναι η γκρίζα ζώνη. τα θέματα που θέλουμε να συζητήσουμε μαζί τους είναι ποια είναι τα περιεχόμενα εκείνα που παραβιάζουν τι τις δικούς τους όρους, their own terms of use και να τους ζητήσουμε από τους ίδιους, όχι από εμά, να τους ζητήσουμε να αποσύρουν το περιεχόμενο εκείνο το οποίο θα εντοπιζόταν από τα κράτη-μέλη και από την Ευρωπόλη, όπως έλεγε και ο Ντεπρέ, ως κάτι παράνομο. Τώρα, όσον αφορά την εκπαίδευση, θα ήθελα να πω ότι η Ευρώπη έχει νέα προγράμματα που διαδέχονται το Εράσμο στο νεολαία και ε, πολίτες. 1,5 δις ευρώ έχουν διατεθεί. Το μεγάλο όφελος είναι ότι δεν είναι προγράμματα τα οποία ε, έχουν την απόχρωση ασφαλείας. Είναι προγράμματα που όπως λέτε πολλοί αφορούν την εκπαίδευση, την πρόληψη, το critical thinking, την κριτική σκέψη, την ανάγνωση των μέσων, ούτως ώστε να, <laughs> εκπαιδεύονται οι νέοι σπουδαστές, η νέα γενιά των πολιτών, να έχουν κριτική σκέψη και να έχουν αντοχέ όσον αφορά την προπαγάνδα. Θα ήθελα να πω και κάτι χρηματοδότηση τη Δημοκρατία. Έχουμε κάτι να προτείνουμε του επόμενου μήνε όσον αφορά το θέμα. Ένα σύστημα παγώματο των περιουσιακών στοιχείων των τρομοκρατών στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, υπάρχει το listing και το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων προβλέπεται από τις αποφάσεις ε, για τρομο, περί τρομοκρατίας Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ. Δεν έχουμε τίποτα ε, εμείς Ευρωπαϊκή, ε, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι παράδοξο. Γραμματικά λοιπόν αναφέρει σημαντικότατα σημεία η έκθεση. Έχουμε δραστηριοποιηθεί από αυτόν. Μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, περισσότερα και ταχύτερα με τη δική σας υποστήριξη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για τώρα η Ρασίδα. Ε, Όντω ακούσαμε πλούσια σχόλια, παρατηρήσει ερωτήματα. Ε, μου μιλήσατε για την ε, ε, προσέγγιση με τη συγκριτική μεθοδολογία, ποσοτική, ποιοτική. Μας μιλήσατε για το Ηνωμένο Βασίλειο. Όντως, ε, πρόληψη και καλέ πρακτικέ Υπάρχουν πολλά καλά παραδείγματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, πληροφορίες, πειράματα γίνονται και ε, σε σχέση με άλλες χώρες ε, μα εντυπωσιάζει η αγαστή συνεργασία των ΟΤΑ με το κράτος. Όλοι εμπλέκονται και στο ισότιμα σε κάποιες άλλες χώρες πάλι υπάρχει μια ιεραρχία ή εν πάση περιπτώσει απαξιώνεται η εργασία κάποιων οργανώσεων σε ορισμένα μέρη. Ε, επίσης, ε, κάποιοι για πολιτικούς λόγους δεν συνεργάζονται με ε, με, μη κυβερνητικέ οργανώσεις ή ενώσεις ή συνδέσμους κτλ. Ενώ ε, ο απότερος στόχος πρέπει να είναι η αποτελεσματικότητα. Ναι, γίνεται δουλειά, υπάρχουν πληροφορίες, υπάρχουν στοιχεία. Με ρωτήσατε για την ποιότητα. ξέρετε, το θέμα είναι η ανάλυση των πληροφοριών. εκεί χωλένει το σύστημα, διότι δεν ξέρω αν είναι ε, πρόσφορη η μέθοδος ανάλυσης που χρησιμοποιείται σε σχέση με τα διαθέσιμα στοιχεία. Ε, για την ερώτηση της Άννα Δίκαιο έχετε, υπάρχει θέμα ορισμού και διατύπωσης. Όταν μου ζητήθηκε να συντάξω την έκθεση, αντιμετώπισα ακριβώς αυτή την δυσκολία, ριζοσβαστικοποίηση, αλλοδαπός μαχητής που δεν είναι όμως αλλοδαπός όλες αυτές οι έννοιες και η έννοια της ριζοσπαστικοποίησης. Μπορεί κάποιος ε, να είναι ριζοσπαστικός και φονταμενταλιστής ε, χωρίς όμως να αναλαμβώ ποτέ τρομοκρατική δράση. Ε, είναι τάτσι το ζήτημα, όπως λέμε. Πολύ λεπτό. Όμως να, ε, δεν θα πρέπει να είμαστε αφελείς. Ε, θα χρειαστούμε ένα καλό ορισμό ακριβώς για να καταλήξουμε και στις αποτελεσματικότερες λύσεις. Όντως θα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένοι στόχοι μας για να βρούμε και τη σωστή διατύπωση. Τι σημαίνει ριζοσπαστικοποιούμε. Όχι ότι θα παριθμίσουμε όλους τους ριζοσπαστικοποιημένους, αλλά ριζοσπαστικοποίηση σημαίνει ε, να κάποιος να έχει διαπράξει μια αξιόπινη πράξη πράξη ή να έχει παρακινήσει κάποιον άλλον να, την ε, να διαπράξει την αξιόπινη πράξη. Αυτά, αυτό ε, συνιστά τη ριζοσβαστικοποίηση και ε, υπάρχουν κάποιες χώρες που έχουν θετήσει αυτόν τον ορισμό, άλλες πάλι όχι. Υπάρχει και κάτι άλλο που δεν πολύ συζητούμε, δεν θυμάμαι ποιο το είπε. Ε, υπάρχει το θέμα της Ισλαμοφοβίας. το Ισλάμ δεν είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι θέμα δημοσίου διαλόγου ε, στην Γαλλία. Ε, η αλητία είναι το ζήτημα, όχι το Ισλάμ. Ε, πρόκειται για αποβράσματα της κοινωνίας που διαπράττουν με αξιόπινες πράξεις χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την θρησκεία αυτό μια θρησκεία είναι. Μπορεί κάποιο να διαθετήσει ή όχι. Λοιπόν, εγώ σας λέω ξεκάθαρα πως ε, σήμερα το να είναι κανείς μηχανικός, ε, πυρηνικός φυσικός ε, ή, ε, και έχει ένα όνομα που θυμίζει Ισλάμ, δυσκολεύεται να βρει δουλειά. Λοιπόν, θα πρέπει να αποναρκοθετήσουμε αυτό αυτή την περιοχή διότι γίνεται ταμπού το ζήτημα τελικά όμως είναι αλληλένδετα αυτά τα θέματα για τη Σαουδική Αραβία δεν θα διαφωνήσουμε αυτή η χώρα Ε, ξέρετε τι ισχύει για την ανισότητα των δύο φύλων, για τα δικαι... την έλλειψη δικαιωμάτων των γυναικών. Υπάρχει ένα πρόβλημα, υπάρχει μια σύγκρουση αξιών με τη δική μας οικογένεια. Εάν θεωρούν κάποιοι ότι είναι μετριοπαθής η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας, τότε έχουμε αξιακό βασικό πρόβλημα. Για τους αλλοδαπούς μαχητές, καλά τα είπατε για τις Ιρακινές αρχές και εγώ ήρθα σε επαφή μαζί τους και μας είπαν «Μα τι αλλοδαπή και κολοκύθια, δική σας ε, υπήκοη ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε θα πρέπει να μας υποστηρίξει για το θέμα των οικογενειών, των οικογενειών συγγνώμη, και του περιβάλλοντος, ε, δηλαδή για την ριζοσπαστικοποίηση ή την ευνίδια αναχώρηση ενός παιδιού μένουν ε, οικογένειες ε, αποσβολωμένες, δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν. Μπορεί κάποιος, όπως σας είπα προηγουμένως, να ριζοσπαστικοποιείται, να γίνεται φόντα χωρίς όμως ποτέ να υποπέσει σε τρομοκρατική δράση. Λοιπόν, χρειαζόμαστε ορισμό, γιατί ούτε πρόληψη ούτε κυρώσει μπορούμε να ε, έχουμε χωρίς ορισμό. Χρειαζόμαστε ορισμό ε, και με τα στατιστικά δεδομένα μπορώ να σας αποδείξω ότι τα θύματα της ριζοσπαστικοποίησης είναι οι μουσουλμάνοι πρώτοι και καλύτεροι, χειρότεροι μάλλον. για την ανταλλαγή πληροφοριών. Καλά τα είπατε. Ε, ο κύριος Κίρκοπ ήρθε ο ίδιος και μας είπε ότι αν ε, ε, θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε τα όπλα που έχουμε στα χέρια μας. Δηλαδή, οι υπηρεσίε πληροφοριών να συνεργαστούν. Για πολιτιστικούς λόγους όμως υπάρχουν κάποιες υπηρεσίε πληροφοριών που δεν θέλουν να συνεργαστούν με άλλες γιατί θεωρούν ότι είναι ευαίσθητα τα δεδομένα και θα πρέπει να επιδιώξουμε μια αυξημένη συνεργασία των υπηρεσιών πληροφορίων. Να, τώρα να αποδίδουμε ε, όλα τα λάθη ε, στο διαδίκτυο. Είπατε ότι δεν είναι καλό. Μα δεν το είπα αυτό. Είπα ότι είναι ένα, μια αιτία ριζοσπαστικοποίησης ε, ε, και ότι ο εικονικός, η εικονική αυτή πλατφόρμα ο, τι συμβαίνει, είναι εκεί, υπάρχουν κάποιοι που δεν είναι ενταγμένοι στην ε, κοινωνία και μέσα από αυτά τα βίντεο που κυκλοφορούν μέσα από τους ιστοτόπους ε, ριζοσπαστικοποιούνται γιατί ξέρετε υπάρχουν, ε, αν δείτε είναι Hollywood τελείως, είναι, το περιγράφουν την, την κατάσταση παραμυθένια και έτσι ε, προσιλητίζουν τους νέους και γυρίζουν απογοητευμένοι γιατί όταν ε, πάνε και βλέπουν τι γίνεται στο Ισλαμικό κράτος, καμία σχέση δεν έχει με το βιντεάκι που τους έδειξαν. Ε, κοιτάξτε, ε, γιατί χρειαζόμαστε μία έκθεση, για να έχουμε μία ε, παγκόσμια ε, συμφερική μάλλον στρατηγική. Αυτή είναι και η ουσία της έκθεσής μου, αλλιώς δεν πρόκειται να καταφέρουμε τίποτα. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος ε, είπε ότι γίνονται σπασμωδικές κινήσεις για τις βέλτιστες πρακτικές. Όχι, υπάρχουν, όμως αυτό πρέπει να κάνουμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να γενικευθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Μπάρβαρα Σπινέλη μας έλεγε για την καταστολή ότι έχει ενδιασμούς για, ως προς το γενικό προσανατολισμό και για τη ριζοσπαστικοποίηση στις ε, φυλακές. Εμεί εστιάζουμε υπερβολικά την προσοχή μας ε, στην καταστολή και αυτό να οδηγήσει τελικά σε διακριτική μεταχείριση μέσα στα σοφρονιστικά ιδρύματα. Όχι το αντίθετο επιδιώκουμε με τα πειράματα που κάνουν και εντάξει καλά τα λέτε ότι στην Ιταλία και στη Γαλλία ε, Είχαμε μεγάλη απομόνωση τότε με τις τρομοκρατικές ομάδες, με τους Βάσκους και τους ε, τους Κορσικανούς ή με τους μαφιόζους ε, στην Ιταλία είχαν απομονωθεί στις φυλακές. Όμως πέραν αυτού μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και όλοι αυτοί που συναναστρέφονται αυτούς τους ανθρώπους και αυτό που χρειαζόμαστε είναι να δούμε τα πρώτα σημάδια, να παίρνουμε τις πληροφορίες, ε, δηλαδή δεν είναι λύση να τους απομονώνουμε, να επιδιώκουμε την πλήρη απομόνωση αυτών των ανθρώπων, έτσι δεν ε, ε, προωθούμε την πρόληψη, ούτε επιδιώκουμε την, το διαχωρισμό, τη διακριτική μεταχείριση αυτών των ανθρώπων. Σχόλια τη κυρία εκτός μικροφώνου. Ε, όχι, υπάρχει ε, ανάμεσα στην απομόνωση και τη διακριτική μεταχείριση κατά κάποιων ομάδων ε, για την πρόληψη υπάρχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, εμεί θέλουμε οι ειδικέ προσεγγίσεις σε σχέση με αυτούς που ε, ριζοσπαστικοποιούνται στις φυλακές. Στη Φρέν, στη Γαλλία, παραδείγματο χάρη, ποια προσέγγιση ε, ακολουθούν ε, όταν βλέπουν ότι κάποιος ριζοσπαστικοποιείται, τον παρακολουθούν στενότεροι για τους ημάμιδες. Ναι, αληθεύει, συμβαίνει αυτό, τους στέλνουν στις φυλακές, αλλά θα σας πει και κάποιος το θέμα δεν είναι ο ημάμ, ο ημάμις. δεν αυτοί που ριζοσπαστικοποιούνται ε, σίγουρα δεν τους προκύπτει από αυτό. Ε, αφήστε που ε, οι χειρότεροι είναι Ευρωπαίοι, δεν μιλούν καν αραβικά και δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε λοιπόν ε, το, το επιχείρημα της γλώσσας. Ε, κυρία Σπινέλη, Ξέρετε, ε, εγώ ε, διαφοροποιούμε λίγο σε σχέση με την ομάδα μου για το PNR. Συζητήσαμε αυτό το θέμα της προστασίας των δεδομένων και της χρήσης των δεδομένων. Αυτό είναι ένα πραγματικό ζήτημα. Έχω όμως και εγώ ερωτηματικά για την ε, χρησιμοποίηση και την προστασία των δεδομένων. Δεν ειναι είναι άσπρο-μαύρο αυτό το ζήτημα, δεν είναι η καλή και η κακή, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να βρίσκουμε και συμβαστικές λύσεις. Η κυρία Λάμπερτ μας μίλησε για την, τον ορισμό ε, της αστικοποίησης. Ε, καλά τα είπατε, μας μιλήσατε για τα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας εκεί δεν μιλάμε για τον ε, ριζοσπαστικό Ισλάμ Χρειαζόμαστε έναν ορισμό, ούτως ώστε να προτείνουμε αποτελεσματικές λύσεις. Θα συμφωνήσω μαζί σας ε, και στο προήμιο, στην εισαγωγική μου παρουσίαση, είπα ότι ε, ο ορισμός θα είναι ε, ένα από τα ουσιαστικότερα ζητήματα, αλλιώς θα έχουμε γενικές κατευθύνες γραμμές που θα είναι άχρηστες. Ε, αποστιγματοποίηση. Συμφωνώ σημαντικό. Η παιδεία είναι μέρος της πρόληψης. Ναι, ναι, αληθεύει. Και για όσους επιστρέφουν πρέπει να τους δώσουμε μία λύση. Δεν μπορεί να είναι μόνο δικαστική η λύση. Έρχονται, επιστρέφουν κάποιοι που δεν έχουν διαπράξει κάποιο έγκλημα. Δεν έχουν διαπράξει ε, καμία αξιόπινη πράξη, όμως ε, έχουν υποστεί κάποιο τραύμα και πρέπει να τους να προβλέψουμε συνοδευτικά μέτα Κάποιοι στην, ε, στο κόμμα μου, στη Γαλλία, λένε ότι ε, ε, πρέπει να απαγορέψουμε την επιστροφή τους. Μα εγώ δεν συμφωνώ Πώς θα βοηθήσουμε αυτά τα άτομα και τις οικογένειές τους, πώς να απαγορέψουμε την επιστροφή τους. Επίσης μας μιλήσατε για τις αιτίες της βαστικοποίησης. Δεν θέλω τώρα να το βλέπω μικροκομματικά το ζήτημα, όπως να λέμε τώρα ότι πρόκειται για ε, προβληματικούς από πλευράς ε, κοινωνικής. Όχι, ξέρετε, εγώ έχω υπηρετήσει και στο δικαστικό σύστημα και μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν κάποιοι που ξεκάθαρα θέλουν να διαβάσουν τρομοκρατικές συνέργειε κατά μιας δυτικής κοινωνίας. Ας μην τα κοινωνικοποιούμε όλα. Υπάρχουν, ναι, υπάρχει ε, η ανάγκη της πρόληψης και των κυρώσεων, όμως υπάρχει το θέμα της ενημέρωσης, της ενσωμάτωσης, της στήριξης των οικογενειών ε, με τα εργαλεία της απορριζοσπαστικοποίησης ε, μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Η καταστολή όμως είναι απαραίτητη ε, για όποιους έχουν διαπράξει μια εγκληματική ενέργεια γιατί έχει αποτρεπτική ισχύ ένα τέτοιο μέτρο, μια τέτοια κύρωση και πιστέψτε με όπως και για την καταπολέμηση της Ισλαμοφοβίας η ποινική κύρωση έχει την ίδια αποτρεπτική ισχύ. Επίσης, κύριε Ντιουπρέ, είπατε ότι ήμουν λίγο αυστηρή. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι μας έρχονται αυτά τα επεξηγηματικά ε, σημειώματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ωραίες αρχές εμείς όμως πρέπει από τα ωραία λόγια να περάσουμε και στη δράση. Ε, καλά τα λόγια, όμως χρειαζόμαστε συγκεκριμένες πράξεις. Για τη Europol. Θα συμφωνήσω μαζί σα. Η Europol όντως μπορεί για το παράνομο περιεχόμενο να δράσει και α, να συνδέσω και ένα άλλο ερώτημα. Μου λέτε είναι λογοκρισία. Ε, όχι, δεν είναι. Είναι παράνομο ή δεν είναι αν ε, δεν είναι παράνομο, είναι, απαγορεύεται απλώς. Δεν πρόκειται για λογοκρισία. Δηλαδή, τα παρά, το παράνομο περιεχόμενο θα πρέπει να απαγορεύεται και αν κάποιος δεν συμφωνεί υπάρχουν ένδικα μέσα. Είναι, ε, υπάρχει κράτος δικαίου, υπάρχουν... Ε, μέσα προσφυγής ε, και ίσως θα έπρεπε να τα αναπτύξουμε περαιτέρω, να τα προωθήσουμε, να τα εγγυηθούμε ή νόμιμο θα είναι ή παράνομο το περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Δεν πρόκειται για ηθική κρίση. Κύριε Ντεπρέ, λέγατε Α, που δεν κάνει τίποτα δεν μπορεί να τον τιμωρήσουμε. Όταν, μετά την όχληση μπορείτε να του πείτε ότι ε, θα πρέπει να αφαιρέσετε το παράνομο περιεχόμενο. Αν δεν το αφαιρέσει τότε ε, παραβιάζει το νόμο και μπορούμε να κινηθούμε δικαστικά. Για ποιο σημείο... Τέλο πάντων θα τα πούμε κατηδίαν αυτά. Πολύ ενδιαφέρουσα η ανταλλαγή απόψεων και συγγνώμη που σας ενοχλώ, λέει ο Πρόεδρος, αλλά περνάει η ώρα. Ναι, ένα λεπτάκι. Ρασίδα, δεν χρειάζεται να απαντήσει σε όλους, ε, Έπρεπε να στο είχα πει εγώ. Μπορεί τώρα να νιώθεις υπόχρη ε, να, ε, απαντήσει σε όλους μέχρι 24. Θα καταθέσετε και τις τροπολογίες τους ε, οι συνάδελφοι. Ξέρεις, ε, ωραίο είναι που απάντησε σε όλους, αλλά ξέρει δεν υποχρεούσε να το κάνεις. αν μπορεί να περάσει σε συμπεράσματα, διότι απάντησε σχεδόν σε όλους. Ναι, μόνο για την Επιτροπή, επειδή μας είπε πω ε, υπάρχουν κάποιε λεπτές χρειές, μα υπάρχουν πολύ λεπτές χρειές μέσα στην έκθεση, για το προπολογισμό του ΡΑΝ του δικτύου, μα χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είναι σημαντική η δράση. Τώρα το να πούμε ότι ε, μπλέκεται και συμμετέχει και ε, mm. το ΝΕΤ είναι όπως σε μία ε, σχέση διαπροσωπική, ε, ερωτική αν θέλετε, χρειάζεται να περάσει κανείς και στην πράξη. Πέρα από τα ωραία λόγια και τις δηλώσεις. Και ε, επίσης ε, για τη χάρτα, εάν δεν υπάρχει εφαρμογή θα πρέπει να δράσουμε και εμείς για την παιδεία. Α, ναι, όχι, ξέρετε για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Ε, λέγαμε για το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων. Λέει η κυρία Γκόμες, να τα παγώσουμε τα περιουσιακά στοιχεία των τρομοκρατών. Ένα αυτό και άλλο να έχουμε την ειχνηλασιμότητα της χρηματοδότησης από πλευρά κράτων μελών προς οργανώσεις, προς σχολεία, θρησκευτικά κτλ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τίποτα δεν έχει γίνει για, το δεύτερο, για τη δεύτερη περίπτωση, για τη χρηματοδότηση από πλευρά κρατών και θα θέλαμε να δραστηριοποιηθεί και σε αυτόν τον τομέα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σίγουρα θα σα υποστηρίξουμε. Παιδεία, έρασμο, ε, το υπόσχομαι θα σταματήσω, Κλοντ. Ε, συγγνώμη, αλλά αυτοί οι νέοι ε, δεν μπορούν να πάνε στο έρασμος, ε, δεν είναι για την κοινωνική του τάξη, είναι για ε, τις μεσαίες και πάνω τάξεις ε, το έρασμος. Ε, οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε για τάξεις που είναι κάτω από τη μεσαία τάξη δεν υπάρχει τέτοια πρόσβαση για ενημερωτικά προγράμματα που θα προωθούσε μέσα στο έρασμος. Δεν μπορεί έτσι να προωθήσει τις αξίες της Ευρώπης, τις αξίες της αλληλεγγύης. Σας ευχαριστούμε κυρία Ρασίδα Ευχαριστώ. Ήταν πληρέστατη η συζήτηση όπως θα έπρεπε. Υπήρξαν και ανησυχίες και έπαινοι. Όποιοι υπήρχαν ανησυχίες για την κατεύθυνση της έκθεσης, εξεφράστησαν, προσπάθησες να απαντήσεις. Όπως έπρεπε έγιναν τα πράγματα. Υποβολή τροπολογιών μέχρι 25 Ιουνίου. Δεν απέχει και πολύ. Παρακαλώ λοιπόν να υποβάλλετε σχετικές τροπολογίες συνάδελφοι και ελπίζω να έχουμε ε, την έκθεση έτοιμη σωστά, προετοιμασμένη. Θέλουμε έγκαιρα να είμαστε έτοιμοι για την ψηφοφορία στις 4 και 20. Θα στριμώξουμε το επόμενο θέμα, είναι το δικό μου ψήφισμα όμως το επόμενο θέμα. Θα το στριμώξω ίδιος, θα το ζουπίξω και θα προχωρήσω γρήγορα. Όπως λέω και στο γραφείο μου έχει αναβληθεί περισσότερο από κάθε άλλη φορά το θέμα αυτό, γιατί είναι το δικό μου. Με κάθε σεβασμό προς εκείνους και προς το πρόσωπό μου, θα προσπαθήσω να το εκτελέσω. Ίσως θα περιορίσουμε τον αριθμό των ε, ομιλητών για να πετύχουμε την προθεσμία, το όριο, το χρονικό των 16 και 20. Να κάνω μια εισαγωγή λοιπόν. Σχέδιο προτάσεως ψηφίσματος ερώτηση για προφορική απάντηση. Υιοθετήθηκε στην Ολομέρεια πέρσι το ψήφισμα μετά από την έρευνα για την ηλεκτρονική παρακολούθηση, μαζική παρακολούθηση. Ήμουν εισηγητή. Μα ανετέθε η συνέχιση τη παρακολούθηση του θέματο και να ξανααναφερθούμε στην Ολομέλεια, στην προηγούμενη ε, θητεία το θέσαμε. Για να το πετύχουμε αυτό λοιπόν, το σκοπό, οι πολιτικέ ομάδε αποφάσισαν να απευθύνουν προφορική ερώτηση προ το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ολομέλεια και να θετήσουν ένα ψήφισμα. Αυτή ήταν η υιοθετηθήσα μεθοδολογία. Σήμερα λοιπόν θα παρουσιάσω όσο πιο γρήγορα γίνεται το κείμενο, σχέδιο κειμένου και μετά θα γίνει μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων. Επιτρέψτε μου συνάδελφοι λοιπόν να σκιαγραφίσω τάχιστα τα βασικά σημεία του σχεδίου προτάσεως ψηφίσματος εν είδη αγωγής. Λοιπόν, στην προηγούμενη θητεία, το λέω για αυτού που δεν ήταν εδώ, η Επιτροπή έκανε έρευνα, δεξιά έρευνα, όσον αφορά τη μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Και υιοθετήσαμε τελικά το ψηφιακό habeas corpus τον Μάρτιο του 2014. Η έρευνα ήταν άνευ προηγουμένου στη φύση τη. 16 ακροάσει διεξήχθησαν και συζητή σε ψηλού επίπεδου με συμμετοχή ευρωγνωμόνων από πλευρά Ευρωπαϊκή Ενώσεω, ΗΠΑ και Βραζιλία. Ακολούθησε ένα ψήφισμα που προσπαθούσε να προβλέψει εξελίξει. Θέλαμε να εξασφαλίσουμε ότι συγκεκριμένε προτάσει θα μπορούσαν να συνεχιστούν και στη νέα θητεία και να, είναι ύψιστη, να έχουν ύψιστη προτεραιότητα στο πρόγραμμα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Παρόλο που στριμώχνουμε το θέμα τώρα, αυτή ήταν η κεντρική ιδέα μα, στη δεύτερη φάση τη έρευνα. Λοιπόν, η Επιτροπή έπρεπε να παρακολουθεί στη διαδικασία και να αναφερθεί σε εσά για τι εξελίξει. Λοιπόν, προθεσμία για τι τροπολογίε είναι 29 Ιουνίου. Αυτή είναι η καταληκτική προθεσμία. Όσον αφορά τη διαδικασία, θέλαμε να ακούσουμε καταρχά τι απόψει Επιτροπή και να ακολουθήσουμε τη διαφανέστερη δυνατή διαδικασία. Γι' αυτό αποφασίσαμε τη συγκεκριμένη διαδικασία. Από την έγκριση της εκθέσεως πέρσι συνεχώς είχαμε εξελίξεις, είχαμε και άλλες αποκαλύψεις από τον Έρβαν Σνόντον για την συλλογή πληροφοριών μέσω αναγνωρίσεως προσώπου, ε, παρεμβολή στους παρόχους τηλεπικοινωνιών, παρακολούθηση εμπιστευτικών συνομιλιών, ε, νομικών ε, και hacking. Και επίσης υπήρξε και παραβίαση των της παραγωγής και των ε, μικρών τσίπ που μπαίνουν στις κάρτες και του μεγαλύτερου παραγωγού τσίπς. Ε, και θέλαμε να δοθεί αποζημίωση ε, όσον αφορά τους πολίτες των οποίων τα δικαιώματα παραβιάστηκαν. Ε, και είχαμε και επίση και το νομοθέτημα των ΥΠΑ όσον αφορά τι βασικέ ελευθερίες. Λοιπόν, το σχέδιο ψηφίσματος παρακολουθεί τις εξελίξει όσον αφορά τι δράσει που προτείνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση για, την Ευρωπαϊκή, για το ψηφιακό habeas corpus. Και θα συνοψίσω λοιπόν τι ζητούμε όσον αφορά του ασφαλείς λιμένες. Υπήρξαν αιτήσει για να ανασταλούν οι ασφαλεί λιμένε και περιμένουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γραπτό να μα δώσει λεπτομέρειε για οποιασδήποτε συμφωνίε που πετέφθη όσον αφορά τι 30 συστάσει που απεστάλησαν στη ΣΥΠΑ. Όπω γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποσχέθη να μα ενημερώσει πέρσι το καλοκαίρι, αλλά η Επιτροπή ακόμα τελεί εν αναμονή και περιμένουμε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να λάβει τι σχετικέ αποφάσει για τι ε, Έχουμε το Συμβούλιο θετεί δευτερογενή νομοθεσία όσον αφορά τους κανονισμούς. Ε, να στηρίξω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα το Κοινοβούλιο δεν πρόκειται να δεχτεί οδήποτε νομοθεσία η οποία εισάγει χαμηλότερε προδιαγραφέ από αυτέ που ήδη ισχύουν λόγω τη οδηγία των 95 και δεύτερον το Συμβούλιο θα πρέπει να προσπαθήσει ούτω ώστε να πετύχει συμφωνία για την οδηγία, την προστασία των δεδομένων και την επιβολή του νόμου μέχρι τον Οκτώβριο του 2015. Αυτέ είναι οι δύο βασικέ στοιχεία, τα δύο βασικά σημεία που ήθελα να τονίσω. Τρίτον, όσον αφορά τη συμφωνία ε, ομπρέλα. Από την υιοθέτηση τη έκθεση, οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να αποζημιώσουν του πολίτε Ευρωπαϊκή Ενώσεω και ήταν βασικό αίτημα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω Καλωσορίζουμε την νομοθεσία του 2015 που θεσπίστηκε όσον αφορά την αποζημίωσή του ε, και την ε, καλωσορίζουμε την έγκριση από το Κογκρέσο. Και τέταρτον, η, μη, αντιδημοκρατικό έλεγχο. Ζητήσαμε από τα Εθνικά Κοινοβούλια να αποκαλύψουν τα συστήματα ελέγχου που έχουν όσον αφορά τι μυστικέ υπηρεσίε και καλέσαμε να παραστούν στη διήμερη διάσκεψη επ' αυτού και ευχαριστώ του συναδέλφου που μπορέσαν να παραστούν. Έγινε Πέμπτη και Παρασκευή, εδώ και μερικέ ημέρε, αυτή η διάσκεψη ε, ήταν πολύ επιτυχής η διάσκεψη και για πρώτη φορά Γερμανία, Ιταλή, Γερμανικό, Ιταλικό, Βελγικό Κοινοβούλιο προσεκλήθη. Τα Εθνικά Κοινοβούλια συζήτησαν και αντάλλαξαν βέλτιστες πρακτικές. Βεβαίως δεν έχουμε εδώ αρμοδιότητα για κάτι τέτοιο, αλλά μπορούμε να ανταλλάξουμε τις βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών και νομίζω ότι αυτό το κάναμε. Λοιπόν, πέμπτον, ε, η ασφάλεια του λογισμικού και των ε, ηλεκτρονικών συστημάτων. Κάναμε συστάσεις στο Συμβούλιο όσον αφορά την αύξηση ασφαλείας ε, της ιδιωτικής ζωής ε, online και τη προστασία των υπολογιστών και του λογισμικού όσον αφορά την ασφάλεια του Κοινοβουλίου. Συνεργαστήκαμε με την κυρία Βάλιαν, τον Κάλο Βαλέλα, τι αρμόδιε υπηρεσίε και δεχτήκαμε τι τελικέ εκθέσει όσον αφορά τι δράσει τη αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Κοινοβουλίου. Ε, διοργανώνει μια σκέψη επιτροπή για την προστασία τη ιδιωτική ζωή στο διαδίκτυο και την αύξηση τη ασφαλεία στο διαδίκτυο και την προστασία του διαδικτύου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θα λάβει τέλο προ το τέλο του 2015. Για αυτά τα δύο σημεία λοιπόν ξανά τίθεται ένα θέμα της δικής μας συστηματικής παρακολούθησης και συνέχειας που θα δώσουμε στο ψήφισμα. Έκτον, όσον αφορά την προστασία των πληροφοριοδοτών, μίας από τις συστάσεις από την προηγούμενη θητεία που συμπεριλαμβάνεται στο ψήφισμα. Ζητήσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξεγάγει μία εξέταση και να κάνει μια επισκόπηση όσον αφορά τη δυνατότητα να υπάρξει ένα πρόγραμμα προστασία των πληροφοριοδοτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι κατήποτε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καλούμε ξανά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τέλο του 2016 το αργότερο να υποβάλει μια σχετική ανακοίνωση. Έβδομον, Όσον αφορά τι τεχνικέ εξελίξει από τι εταιρείε ε, του οικισμικού, δίνει το ψήφισμα λεπτομέρειε όσον αφορά τι αντιδράσει από εμπορικέ εταιρείε όσον αφορά την κρυπτογράφηση και την μετακίνηση των διαφόρων υπολογιστικών εφών και ανακοίνωση διάφορε εταιρείε, ώστε τελικά να υπάρχει τελική κρυπτογράφηση ε, και να αποφευθεί έτσι η μαζική παρακολούθηση και φτάνω στο τέλο σχεδόν. Βλέπουμε από την όλη κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Χάμπεας Κόρπους ότι πόρα απέχουμε από την εκπλήρωση όλων των συστάσεων μας σε επίπεδο κρατών μελών έγιναν περισσότερε συζητήσει και ευαισθητοποίηση, περισσότερο ποτέ όσον αφορά τα θέματα τη προστασία ιδιωτική ζωή, όμω αυτό δεν ε, ακολουθήθηκε από συγκεκριμένα μέτρα. Περιορισμοί από τι μονάδε επιβολή του νόμου και τι αστικέ υπηρεσίε δεν ευθυγραμμίστηκαν με το ψήφισμα και θεώρησαν ότι οι δραστηριότητέ του είναι χρήσιμε και ότι αντιδρούν κατά ε, πρωτοβουλειών, προσπαθούν να κάνουν τι επικοινωνίε ασφαλέστερε και πρέπει να μα βοηθήσουν για την κρυπτογράφηση, για την προστασία. Δεν θέλουν να μα βοηθήσουν για την κρυπτογράφηση, για την προστασία του ατόμου. Στο ψηφίσμά μα έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να πάρουμε και κρίνοντας πρέπει να πω ότι ήμουν ιδιαίτερα προκλητικός προτείνοντα ότι όσον αφορά το ψήφισμα έχουμε ακόμα κενά. Θα ήθελα να πω ότι έχουμε κενά και δώσω τα, το λόγο στα μέλη που παρακολουθούσαν λεπτομερώς το θέμα να ζητήσω ποιες είναι οι απόψεις τους κυρίως τη Ομάδα Παρακολούθηση Monitoring Group. Ο Άξελ Βο είναι ο πρώτος απαραίτητο λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα και για το ψήφισμα να τοποθετηθώ. Περιορίζω, περιορίζομαι όμως λόγω χρόνου σε έξι σημεία. Αφενό στην παράγραφο 4, στο εδάφιο 4 που αναφέρεται και που νομίζω είναι κάπως ανεδαφική πλέον. Μια και εχθές στο Συμβούλιο ολοκλήρωσε τα θέματα της προστασίας δεδομένων και έτσι νομίζω έχει ξεπεραστεί πλέον αυτό το εδάφιο. Εδάφιο 6, παράγραφος 6. Θα έλεγα <clears throat> μετά από αυτά τα οποία γνωρίζουμε μετά από ένα έτος, μετά από αυτό με την δέσμη μέτρων, με αυτόν τον άκαμπτο τρόπο δεν έχει μεγάλο νόημα πια. Μπορεί κανείς ε, παράλληλα να δει κανεί μια εξέλιξη. Αλλά αν τώρα θα πρέπει να θα υπάρξει ολοκλήρωση, τερματισμό, δεν νομίζω πρέπει να εμείνουμε. Πρέπει να υπάρχει ελαστική αντιμετώπιση των πραγμάτων σε σχέση με αυτό το εδάφιο. Παράγραφη εδάφια 9-13 για ασφαλή λιμένα. Έχω την εντύπωση, δεν πρέπει να επαναλάβουμε πάλι εδώ αυτά τα οποία αναφέραμε πέρυσι θα πρέπει να προσαρμοστούμε στα δεδομένα και να πούμε μάλιστα εντάξει υποστηρίζουμε αφενός τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσουμε στη συνέχεια τα αποτελέσματα και θα δούμε όμως ποιες λύσεις και οδούς μπορούμε να ακολουθήσουμε ώστε η αρχή του ασφαλούς λιμένα αλλού ή με άλλο τρόπο να μπορέσει να εφαρμοστεί και τότε μόνο να μπορέσουμε να μεταβούμε αν όλα αυτά δεν λειτουργήσουν και δεν εγκατασταθούν να έχουμε την άρση, την κατάργηση του ασφαλούς λιμένα στο εδάφιο στην παράγραφο 17. Πιστεύω απλά ότι η εθνική ασφάλεια είναι θέμα των κρατών μελών. Και εδώ δεν μπορούμε εμείς ε, να ε, αναλάβουμε αρμοδιότητες, ε, διότι δεν είναι δική μας αρμοδιότητα αυτά τα θέματα. Στο εδάφιο 20 για την TTIP, Συμφωνία Εμπορικών Συναλλαγών και Επενδύσεων, δεν έχουμε κάποια τεκμήρια ότι υπήρξαν κάποιες ε, καταχρήσεις. Γιατί τώρα θέλουμε όλα αυτά να τα καταργήσουμε, δεν μπορώ να το κατανοήσω. Στην παράγραφο 24 τώρα και εδώ έχω την εντύπωση πάλι ότι δεν έχουμε αρμοδιότητες αυτά τα θέματα στο ευρωπαϊκό επίπεδο να τα εγγράψουμε και να τους δώσουμε συνέχεια. Στην παράγραφο 30 θέλω να επισημάνω <clears throat> ότι είναι αυτό το χρονικό πλαίσιο από πλευρά έτους βέβαια αλλά θα έλεγα να μεταθέσουμε το κέντρο βάρους και να πούμε να το κάνουμε αυτό όταν θα είναι αναγκαίο και πρέπει να γίνει και όχι με ένα άκαμπτο χρονικό πλαίσιο. Συνάδελφοι, θα κλείσω με την Εύα Ζολή, την Μπάρμπαρα Σπινέλη, τον κύριο Χόπερ, τον κύριο Κοέλιο, Έρνστ και μπήκε σύμβολη τον κατάλογο των ομιλήτων αν συμφωνείτε. Μην καθυστερείτε. Εντάξει, εγώ φταίω, δεν τα έκανα καλά, αλλά πρέπει να ψηφίσουμε στις και 20. Οπότε παρακαλώ λίγη αυτοσυγκράτηση. Εύα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα, διότι είναι εξαιρετικά ποιοτική η έκθεσή σας και θα την υποστηρίξουμε εμείς οι πράσινοι. Όπως και εσείς. Λυπούμεθα που για το Safe Harbor και για το SWIFT ε, οι συμφωνίες ε, δεν ε, τηρήθηκαν και βλέπουμε ότι συνεχίζεται η μαζική παρακολούθηση των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, όχι μόνο δεν έχει σταματήσει η μαζική παρακολούθηση σε συνεργασία με την NSA και το headquarters στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά παρατηρούμε πως στις περισσότερες χώρες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει και παρακολούθηση από πλευράς της Γερμανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για λογαριασμό των, Αμερικανική Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Είναι σοκ αυτό και δεν ε, είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα η αποκάλυψη αυτή στην κοινή γνώμη. Ε, όπως ε, αναμέναμε. 50 ε, διαφορετικές περιπτώσεις ε, παρακολούθησης είχαμε από πλευρά της Γερμανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Το ίδιο έγινε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι απίστευτο. Επίση, η κατάσταση των συστημάτων πληροφορική, η επίθεση, η κυβερνοεπίθεση που έγινε στην Γερμανική Βουλή. Μα εξοργίζει που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι πιο επίγον να προωθήσει την οδηγία για τι εμπιστευτικέ πληροφορίες που δεν ζητάει κανένα έτσι, πέρα από του λομπίστε, παρά ε, να προωθήσει μια οδηγία για την ενεργοποίηση του μηχανισμού για τέτοιε επίγουσε περιπτώσει. 300.000 πολίτες σε διάστημα μικρότερο από 30 ημέρες ε, το ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ζήτησαν να προωθηθεί οδηγία για το whistleblower και ανταυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την οδηγία για τις εμπιστευτικές πληροφορίες. Ε, Πρόεδρε, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να μιλήσω αλλά δύο λεπτά, διότι υπάρχει και η ανησυχητική νομοθεσία για την υπηρεσία πληροφοριών στη Γαλλία. Χάρη σε αυτή τη νομοθεσία μπορούν να παρακολουθούνται όλοι οι πολίτες χωρίς κανένα δικαστικό έλεγχο. Γιατί λέω χωρίς έλεγχο, διότι είναι γελίο ο δικαστικός μηχανισμός. Ε, υπάρχουν εκατομμύρια ε, υποκλοπών και έχουν τρει που δεν, καν, δεν δουλεύουν καν ε, σε πλήρη απασχόληση. Εύα, ε, θα γίνει ξεχωριστή συζήτηση για το θέμα αυτής του γαλλικού νομοσχέδιου. Καλώ λίγη πειθαρχία, συναδελφοί, γιατί πλησιάζει η ψηφοφορία και μετά πρέπει να φύγουμε και από εδώ γιατί έχουμε την κοινή ακρόαση με τη ΣΕΝΤΕ. Παρακαλώ πειθαρχία, λοιπόν, γιατί έχουμε την ψηφοφορία και την κοινή ακρόαση. Ο κύριος Κύρκο. είμαι πάρα πολύ και ε, εστιασμένος, Πρόεδρε. Όπως μόλις ακούσαμε από την Εύα Ζολή, όχι, όχι, από τον κύριο Βος, Φως, ε, Βάσει του άρθρου 4 παραμένει αυτό εθνική αρμοδιότητα και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σέβεται την εδαφική ακαιρεότητα, τη διατήρηξη της ε, δημόσιας ε, ασφάλειας και βλέπουμε ότι αυτό συνιστά ε, αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών και θα το υποστηρίξω επίσης. Θέλω να υπάρχουν ισχυρές πολιτικές προστασίας των δεδομένων και επίσης τήρηση των νομίμων διαδικασιών από τις υπηρεσίες πληροφοριών. Όμως ε, θα πρέπει να έχουμε ε, εθνικά ελεγκτικά όργανα για την παρακολούθηση της δράσης των ε, υπηρεσιών πληροφοριών. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν έχω κρύψει ποτέ ότι είμαι κατά του, της λειτουργίας του whistleblower ο κύριος Σνόντεν είναι φυγάς ε, κατά τη γνώμη μου και ε, θα πρέπει να επιστρέψει και να δικαστεί στη ΣΥΠΑ. Δεν το έκρυψα ποτέ και ε, ξέρετε, Πρόεδρε, τις τελευταίες δύο ημέρες τι ζημιά έχει κάνει ο κύριος Σνόντεν Στι υπηρεσίες πληροφοριών ε, τον ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου και ε, γενικότερα για τη δυτική ασφάλεια και μπορεί, ε, θέτει σε κίνδυνο εκατομμύρια ζωέ και ίσως έχουν χαθεί και ζωές στην Ευρώπη. Εντάξει, εκείνοι μπορούν να γελάνε για αυτά που λέγεται ο Σνόντεν, όμως εγώ μιλάω για διάσωση ζώνης δεν είναι ανεύθυνο να ε, στέλνουμε την ισχύ διεθνών συμβάσεων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ούτε η ομάδα μου ούτε εγώ ίδιο να το υποστηρίξουμε. Σα ευχαριστούμε. Μπάρμπαρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω, είναι έξοχη η έκθεση και εκφράζεται και σε μία που δεν σας ικανοποιούν και εκφράζεται και προθυμία να προσφύγεται στη νομοθεσία όσον αφορά την μη κινητοποίηση, επαρκή κινητοποίηση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους whistleblowers τώρα, τους πληροφοριοδότες. Δυστυχώς δεν πήραμε σαφείς απαντήσεις και το θεωρώ σοβαρότατο αυτό. Θεωρώ σοβαρότατο να κατηγορεί το Σνόντερ ότι έβλαψε άτομα, κάτι που δεν έκανε. Και ήθελα να ρωτήσω αν είναι δυνατό να συμπεριληφθεί στην έκθεση και η προστασία των δημοσιογράφων πληροφοριοδοτών. Όχι μόνο των εργαζομένων στην εταιρεία, αλλά του πληροφοριοδότη δημοσιογράφου που καλείται να διατηρήσει την, ε, τον εμπιστευτικό χαρακτήρα πληροφοριών που αφορούν τις μεγάλες πολυεθνικές. Έχουμε την οδηγία ε, για το μυστικό των επιχειρήσεων που άπτεται αυτών των ζητημάτων. Αυτά είχα να πω και ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μπάρμπαρα. Καλώς. Καλώς Κοέλιο. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θα ήθελα Πρώτα απ' όλα να σας συγχαρώ Πρόεδρε για το κείμενο που μας παρουσιάζετε και που είναι μια εξαιρετική βάση εργασίας. Μπορεί να βελτιωθεί, όμως κυρίως επισημαίνει όλους τους τομείς που αναφέρεις και που πρέπει να δώσουμε απαντήσεις σε αυτούς. Η μεγάλη μου επιφύλαξη σε σχέση με αυτό το ζήτημα της ε, ηλεκτρονικής παρακολούθησης, μαζικής ηλεκτρονικής παρακολούθησης, είναι ότι αντιδρούμε όταν υπάρχει κάποιο σκάνδαλο μετά από δημοσιεύματα ε, στον τύπο. Το γεγονός ότι ε, επήρε και αντιμετώπισε με το δικό του τρόπο ο Κλοντ Μωράης ε, διασφαλίζει ότι θα είναι θέμα της ΛΥΜΠΕ και δεν θα το ξεχάσουμε αυτό στη δράση μας. Θέλω να υπογραμμίσω δύο πράγματα. Δύο πράγματα. Πρέπει να είμαστε σαφείς στη σχέση μας με τρίτα κράτη. Και δεύτερον, δεν μπορούμε να μείνουμε αδρανείς με την ιδέα ότι αυτό δεν είναι λέει δική μας αρμοδιότητα. Αληθεύει ότι η αρμοδιότητα παρακολούθησης των ε, μυστικών υπηρεσιών είναι εθνική αρμοδιότητα. Όμως αληθεύει εξίσου ότι μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς ε, να ε, εφαρμόζονται οι βέλτιστες πρακτικές. Το παράδειγμα είναι η ακρόαση που διοργάνωσε αυτή η Κοινοβουλευτική Επιτροπή με τους Προέδρους των Επιτροπών των Εθνικών Κοινοβουλίων αρμοδίων για τον έλεγχο των υπηρεσιών, μυστικών υπηρεσιών. Και αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα. Με βάση αυτές τις εμπειρίες και αυτά τα βιώματα μπορούμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο να γνωρίζουμε, να δώσουμε τις σωστές απαντήσεις. Αυτός είναι ο στόχος. Αν σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν λειτουργεί ο κοινοβουλευτικός έλεγχος και δεν υπάρχει δικαστικός έλεγχος, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει υπάρχει κίνδυνος παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Και όταν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, αυτό σίγουρα είναι αρμοδιότητα την οποία δεν μπορούμε να απεμπολίσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Κάρλος. Κορνίλια Ευχαριστώ, Κλοντ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να διαπιστώσω ότι είναι καλό να έχουμε ένα τέτοιο ψήφισμα το οποίο ξανακατατίθεται. Μια και βρισκόμαστε ε, σε ένα τοπίο που έχει αποτελματωθεί και δεν έχει αλλάξει τίποτα και σε σχέση με μυστικές υπηρεσίες όπως γνωρίζουμε συνεχίζουν αυτές τις δραστηριότητες. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης είναι πολύ δύσκολο εγχείρημα. Ακούγεται ωραίο αυτό σε αυτό το ψήφισμα αλλά δεν έχω τέτοια εμπιστοσύνη εγώ. Δεύτερο σημείο, οι δέσμοι μέτρων για τα δεδομένα πρέπει να παραμείνει σε ένα κοινό πλαίσιο. Έχω τη μεγάλη επιφύλαξη κάποια από αυτά τα θέματα μέσα σε αυτήν την οδηγία να αγνοηθεί και να καταποντιστεί. Και στη συζήτηση αυτών των πραγμάτων δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα μπορέσουν να τεμαχιστούν αυτά τα θέματα. Το safe harbor, ο ασφαλής λιμένας, δεν αλλάζει καθόλου τα πράγματα. Μπορούμε λοιπόν να παραμείνουμε σε σχέση με την κατάργηση την οποία είχαμε συστήσει μια και η σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ανταποκρίνεται πλήρως στα αιτήματά μας. Δημοκρατικός έλεγχος είναι, ας το πω έτσι, το ευαίσθητο, η ευαίσθητη κοιλίδα αυτού του προβλήματος συνολικά για τις μυστικές υπηρεσίες. Διαπιστώνουμε επανειλημμένα ότι είναι απόλυτα σε αυτές οι διατάξεις και το είδαμε κατ' επανάληψη. Εδώ πρέπει αυτά να αναφέρονται στα ψήφισμα και να προσαρμόζονται. Πληροφοριοδότες, whistleblowers, είναι έκφραση του, της δημοκρατίας. Δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε αυτούς τους πληροφοριοδότες. Είναι στοιχείο της ελευθερίας και της, έκφρασης, της, της ελευθερίας έκφρασης. Δεν μπορούμε λοιπόν να ακολουθήσουμε μέτρα καταστολής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κορνίλια. Τέλος, Birgit. Ευχαριστώ. Μπορούν όλοι να σταματήσουν τα πηγαδάκια. Παρακαλώ. Καλά, και τι να μην θα το κάνει, ναι, λέω πρόεδρος, ξέρω ότι είσαι φιλόδοξη, αλλά να είστε και ρεαλίστρια ξέρετε θέλω να πω κάτι για την ε, συζήτηση, διότι υποστηρίζω την έκθεσή σας. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω, να επαναλαμβάνω τα ίδια και τα ίδια, όμως ε, όσο δεν αλλάζει κάτι θα πρέπει να θυμίζουμε τι ζητήσαμε στην αρχική έκθεση ε, για την NSA. Δεύτερον, για την εθνική ασφάλεια δεν Έχω μόνο την εντύπωση ότι είναι θέμα δικής μας αρμοδιότητας. Σε πολιτικούς πώς είμαι επιβεβαισμένη ότι πρόκειται για ενωσιακή αρμοδιότητα. Όταν πρόκειται για σοβαρό διασυνοριακό κυβερνό, ασφάλεια, τρομοκρατία, όλα αυτά ε, συνδέονται με ευρωπαϊκές αρμοδιότητες και άρα θα έπρεπε να δώσουμε και μια ευρωπαϊκή απάντηση. για τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών δεν μου αρέσει αλλά τι να κάνουμε υπάρχει. Στην έκθεση της NSA μιλήσαμε για τη Βρετανική Υπηρεσία Πληροφοριών, τώρα μιλάμε για τη Γερμανική Υπηρεσία Πληροφοριών και σχάτως για τη Γαλλική. Ε, πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα στην Ευρώπη για την προστασία των δεδομένων και το πακέτο ζήτω. Συγγνώμη, αλλά χρειαζόμαστε προσέγγιση, διότι αλλιώ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρχει το ίδιο επίπεδο στον κανονισμό και στην οδηγία. Άρα θα συμφωνήσω. Πρόεδρε, με εσά ανακουφίζομαι, λέει ο πρόεδρο, που συμφωνείτε μαζί μου. Ε, όπως ακούσαμε και τον Άξελ Βος, ε, ε όντως ε, δεν θα έπρεπε να ε, διεκπεραιώνουμε έτσι ένα ε, τέτοιο, μια τέτοια περίπλοκη πρόταση. Η προθεσμία 29 χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο, αλλά ξέρετε ε, κάποιες αποφάσεις πρέπει να λαμβάνουμε σε αυτή την Επιτροπή και εστιάσαμε στην προηγούμενη έκθεση. Ε, δεν θα απαντήσω τώρα σε όλες τις ερωτήσεις. Στείλτε τα Μπάρμπαρα στο γραφείο μου και θα προσπαθήσω να σας απαντήσω. Μέχρι τις 29 παρακαλώ οι τροπολογίες. Τώρα πρέπει. Έφτασε η ώρα για την ψηφοφορία. Για ένα λεπτό θα διακόψουμε. Γιατί θέλει να με ενημερώσει για κάποια ζητήματα η γραμματεία. Ξέρω ότι με παρακολουθείτε όλοι. Ένα λεπτάκι λοιπόν ε, διακοπή. Απλώς ε, φροντίστε να έχετε την, ε, τις κάρτες σας. Ένα λεπτό.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 the draft amending budget number 5 2015 of the EU. Λοιπόν, ε, περνάμε στην ψηφοφορία για τον ε, ε, σχέδιο τροποποιητικού προπολογισμού 5 2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 τροπολογία να υπέρ. Mm. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική ένα υπέρ. Κατά. Mm. Αποχές απορρίπτεται, έτσι δεν είναι. check compromise amendment. Έλεγχος για τη συμβαστική 1, παρακαλώ. The vote is closed. Τέρας. Do you want to push your card in because mine wasn't. Συγγνώμη, αλλά δεν λειτουργεί η κάρτα σας.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 compromise one is adopted. Amendment four. Who's for? Ε, η τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται, διόρθωνα πρόεδρο, συγγνώμη. Ε, άρχεται για την τροπολογία 4, ναι, επαλήθευση. Λοιπόν, ξανά. Τροπολογία 3, υπέρ. Κάτα. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6, υπέρ. Κάτα. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5, υπέρ. Κάτα. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος. Άρχεται. Για την τροπολογία 5. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος. Άρχεται η τροπολογία 9. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μπορείτε να σκόνετε και τα χέρια. Για τη συμβαστική 2 τώρα ηλεκτρονικός έλεγχος. That's Εγκρίθηκε. Μπορείτε να σηκώνετε και τα χέρια σας παρακαλώ. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Α, πρώτο τμήμα για την 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. νομίζω χρειάζεται επαλήθευση. Για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 21 παρακαλώ. Πέρασε. απορρίφθηκε. Τροπολογία 22 πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 22. Όχι, για το πρώτο. Τροπολογία 22. Πρώτο τμήμα. Άρχιτη ψηφοφορία. Μέχρι τις 16 22. Ναι. Πρώτο τμήμα. Ε, Παρακαλώ, ψηφίστε για τροπολογία 22, πρώτο τμήμα. Πέρας. Εγκρίνεται. 22 δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται όχι εγκρίθηκε 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Για τελική ψηφοφορία. Παρακαλώ. Τσίπρας. Πέρας. Congratulations, Mr. we have to move to room number... πρέπει να πάμε. Πού πρέπει να πάμε? Colleagues, we move to room number 1E2. E Αίθουσα 1 ή 2. 1 ή 2 για την κοινή συνεδρίαση Λίμπε Σέντερ για την εφαρμογή της